Good morning, ladies and gentlemen. Καλημέρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Να ξεκινήσουμε την ε, κοινή μας δημόσια ακρόαση της Επιτροπής μας και της Επιτροπής γιουρι, Να καλωσορίσω και τον ε, Πρόεδρο Σβόποντα. Θα δώσω το λόγο αμέσως στον Συμπρόεδρο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε Λάνιεν, καλώς ήρθατε αγαπητοί συνάδελφοι και ευχαριστούμε την Επιτροπή σας που δέχτηκε να κάνουμε αυτή την ε, κοινή ακρόαση για το θέμα αυτό. Θα επικεντρωθούμε στην προστασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο των καταγγελόντων είναι πραγματικά σημαντικέ οι καταγγελίε σε μια καλώ λειτουργούσα δημοκρατία. Η Επιτροπή Γιούρη και ο συγητή μα, η συγγητριά μα μάλλον, η κυρία Ροζιέ, βρίσκονται στη διαδικασία να συντάξουν μια έκθεση ε, ίδια πρωτοβουλία για την προστασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο των καταγγελόντων. Οπότε τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνουμε αυτή την ακρόαση. Και τώρα ξαναδίνω την Προεδρία στον κύριο Λάκη. Ευχαριστώ πολύ. Να αλλάξω στην μετρική μου. Έχουμε μετάφραση σε όλες τις γλώσσες. Επίσης υπάρχει web streaming της ε, ακρόασης. Να σας θυμίσω ότι ο κύριε Πρόεδρε, ότι ε, την προστασία των καταγγελόντων ε, την προωθούμε από κοινού. Είναι στην σε διάταξη των επιτροπών μας και Χαιρόμαστε πολύ που και η δική σα ε, Μητροεπή θα κάνει αυτή την έκθεση ίδια πρωτοβουλία. Θα ασχοληθούμε λοιπόν και με την ε, γνωμοδότηση τη κυρία Ροζιέ. Έχουμε τον κύριο Κόφορτ και ε, τον, και δεύτερο συνεισηγητή από τη δική μα επιτροπή. Βλέπω και τρει αντιπροέδρου τη Επιτροπή Πάνα. Δεν είμαστε πολλοί, αλλά οι πιο σημαντικοί είμαστε εδώ. Καλώ ορίσατε λοιπόν και χαίρομαι που έχουμε σήμερα εδώ ε, μια σειρά εμπειρογνωμόνων και όπως πάντα συζητούμε την ε, εκπροσώπηση των γυναικών στα διάφορα βήματα. Έχουμε 35,8 θηλυκά μέλη. Σήμερα έχουμε 5 γυναίκες εμπειρογνώμονες όμως. 100% επιτυχία σήμερα. Είναι πολύ χαρούμενη ημέρα λοιπόν. Καλώς ήρθατε κυρίες. Να σας καλωσορίσω μία-μία, Βιτσιλέντσα Αμπάτσι, βοηθό καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Μάστρικ, η Σαρλότ Γκράς, επικεφαλή του, ε, της μονάδας ανταγωνισμού και συμμόρφωσης του, της ομάδας βαλούρε, η, και Κάθη Τζέιμς, εκτελεστική διευθύντρια του Public Concerns at Work, η Φρεντερίκ Μπεγό, καθηγήτρια στο Κολέγιο της Ευρώπης. Καλώς ήρθατε και εσείς και η Ροζίτα Χαϊκή από εδώ, στην από εδώ πλευρά, ε, επικεφαλής των ε, στρατηγικών ερευνών στο γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολογητή. Σας ευχαριστώ όλες που είστε παρούσες. Συνήθως για κάθε ε, ομιλητή δίνουμε 7 λεπτά για κάποια εισαγωγικά σχόλια. Οπότε θα σας ευχαριστήσω ήδη και για τα γραπτά σας σχόλια. Τα έχουμε και αυτά στο φακέλους μας. Και να ξεκινήσω με την κυρία Αμπάτση. Ε, yes, perfect. Ε, members, dear members of the committee, Αγαπητά μέλη της Επιτροπής, καλημέρα σας και ευχαριστώ που με καλέσατε να συζητήσω σήμερα μαζί σας τους κανόνες που υπάρχουν για τους καταγγέλλοντες στα Ευρωπαϊκά κράτη-μέλη. Η σύντομη παρουσίασή μου έχει τρία, μέλη, τρία μέρη. Καταρχά, θα μιλήσω για την γενική εικόνα, για το ποια είναι η γενική κατάσταση στα κράτη-μέλη, σχετικά με του κανόνε που διέπουν του καταγγέλλοντε. Μετά θα μπω σε λίγο περισσότερε λεπτομέρειε για τα διάφορα στοιχεία των νομικών πλαισίων. Και τέλο, θα δούμε τι προκλήσει και πώ πρέπει να τι αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Το βασικό λοιπόν μήνυμα που θα ήθελα να σας παρουσιάσω είναι ότι Έχουμε μια ε, ένα κατακαιρματισμένο πλαίσιο προστασίας των καταγγελόντων στην Ευρώπη και αυτό είναι πραγματικά πολυεπίπεδο. Τι σημαίνει. Το πρώτο επίπεδο κατακαιρματισμού είναι ότι γενικώ μας λείπουν, ε, μας λείπουν δυνατότητες προστασίας των ε, καταγγελόντων. Δεν έχουν όλα τα κρατημέλη δυνατότητες προστασίας τους και κάποια κρατημέλη έχουν μερικούς κανόνες. Αυτό τι σημαίνει. Ότι αναφέρονται στο, είτε στο ποινικό του δίκαιο είτε στην, ε, στο αστικό για την ε, διαφθορά κτλ. Αλλά δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνε που να αφορούν αμοιβώ του ε, καταγγέλλοντε. Α πούμε, για να δείτε λίγο περισσότερο τι ακριβώ εννοώ, όπως βλέπετε στη διαφανή, η πλειοψηφία των κρατών μελών, 13 συγκεκριμένα, και μπορείτε να δείτε και ποια είναι τα κράτη-μέλη αυτά, παρέχουν μερι, μερικούς ε, κανόνες και κάποια δεν έχουν καθόλου κανόνες ή έχουν πολύ περιορισμένες ε, διατάξεις για την προστασία. Τώρα, όταν, θα, όταν μιλάμε για την εφαρμογή των κανόνων αυτών, ένα κράτος μέλος επειδή έχει νομοθεσία, δεν σημαίνει αυτό κατά ανάγκη ότι και στην πράξη παρέχεται πλήρης προστασία στους καταγγέλλοντες. Οπότε, νομικός, βλέπουμε ότι υπάρχει κάποια βελτίωση. Και αυτό είναι τα, τα καλά νέα. Τα τελευταία δύο χρόνια είδαμε ότι υπάρχει αύξηση και διεύρυνση τη προστασία των καταγγελόντων στα κράτη-μέλη. Α πούμε, είδαμε διεύρυνση τη προστασία στη Γαλλία, στη Σουηδία το 2016 και 2017. Είδαμε νέα νομοθεσία να προκύπτει σε χώρε όπω η Σλοβακία. Γίνονται συζητήσει επίση και στην Τσεχία σχετικά, στην Ισπανία για νέε διατάξει για την προστασία των καταγγελόντων. Οπότε η γενική τάση είναι να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι κανόνε για του καταγγέλλοντε και η νομική προστασία για αυτού να αποτελεί συγκεκριμένο κομμάτι εντό τη νομοθεσία των κρατών μελών. Παρ' όλα αυτά, αυτό που βλέπουμε στην πράξη, και εδώ είναι το δεύτερο επίπεδο της, ε, του κατακριματισμού για το οποίο σα μιλώ, είναι ότι οι κανόνε για του καταγγέλλοντε έχουν πολύ περιορισμένο πεδίο εφαρμογή. Αυτό σημαίνει ότι οι κανόνε, όπω στη Ρουμανία, που έχει πολύ καλή ε, νομοθεσία μεν, αλλά ε, αφορά μόνο στον δημόσιο τομέα δε. Ναι. Οπότε αφήνει έξω με ένα μεγάλο κομμάτι τη κοινωνία. Οπότε αφήνει ουσιαστικά απροστάτευτο του καταγγέλλοντε. Επίση έχει πολύ περιορισμένου τομεί που καλύπτονται. Υπάρχουν κράτη-μέλη που καλύπτουν του ε, ε καταγγέλλοντε όταν μιλάμε για θέματα οικονομικά ή διαφθορά. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει, δεν συμβαίνει γενικώ. Από την πράξη λοιπόν βλέπουμε ότι οι καταγγελίες ε, γίνονται ε, σε, σε ε, υποθέσεις περιβάλλοντος ή υγείας, οπότε όταν υπάρχει τέτοιο είδος κατακαιρματισμού, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει νομοθεσία ή όχι, ακόμη και αν υπάρχει νομοθεσία, τι καλύπτει. Αυτό είναι άλλο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη. Βεβαίω υπάρχουν και καλά παραδείγματα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να τα δείτε στη διαφάνεια, αλλά η Ιρλανδία ας πούμε, και το Ηνωμένο Βασίλειο ξέρω ότι έχουν ε, δημο, ε, πράξεις ε, δημόσιας δημοσίευσης που δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένους κανόνες, οπότε ε, προστατεύεται η δημοσίευση τέτοιων στοιχείων γενικώ. Επίσης, κάποια στοιχεία τώρα. Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, θα επικεντρωθώ σε, μια από τις πιο σημαντικές συζητήσεις, που είναι οι, οι τρόποι με τους οποίους υποβάλλονται αυτές οι ε, εκθέσεις. Για να υπάρχει λοιπόν νομική ασφάλεια για τους καταγγέλλοντες και να έχουμε πραγματική λογοδοσία που θα απορρεύσει από αυτή την καταγγελία, πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα ε, κανάλια ε, για την παρουσίαση αυτών των πληροφοριών. Αυτό που βλέπουμε γενικώ ω τάση είναι ότι τα κράτη-μέλη ε, θεωρούν υποχρέωση των καταγγελόντων καταρχάς να ε, κάνουν την καταγγελία εντός του ε, χώρου εργασία τους, στον εργοδότη του, α πούμε. Αυτό είναι καλό γιατί είναι πολύ κοντά στην πηγή του προβλήματος, αλλά στην πράξη βλέπουμε ότι μπορεί να είναι και αντιπαραγωγικό κάποιε φορέ γιατί ο καταγγέλων ήδη αντιμετωπίζει τις αρνητικές συνέπειες των πράξεών του για αντίπεινα ή για υποβάθμιση της θέσης τους ε, οπότε πρέπει να γίνει μια γενική εποπτεία, μια γενική έρευνα, αξιολόγηση των, ε, της καταγγελίας ε, ή της παράβασης καθήκοντος ή τέλος πάντων της παράνομης πράξης. Επίσης υπάρχουν κάποια επίπεδα καταγγελίας που δεν είναι μόνο εσωτερικά του χώρου εργασίας αλλά υπάρχουν και αρμόδιες αρχές ή και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπό το φως και των συζητήσεων που γίνονται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα έπρεπε να ξανασκεφτούμε λίγο αυτή την υποχρέωση και ίσω να ακολουθήσουμε το παράδειγμα τη Ιρλανδίας, που από τη μία μεν απαιτεί ο καταγγέλων να κάνει την καταγγελία του εσωτερικά, αλλά υπάρχει και σαφ... υπάρχουν και σαφεί εξαιρέσει σε αυτό, που σημαίνει ότι σε περιπτώσει όπου ο καταγγέλων φοβάται ότι μπορεί να υπάρξουν αντίπεινα ή ότι δεν θα υπάρξει κάποια συγκεκριμένη δράση, ο καταγγέλων επιτρέπεται να πάει ε, να κάνει την καταγγελία του σε μια άλλη εξωτερική αρχή ή στα ΜΜΕ. Και βλέπουμε παρόμοια παραδείγματα και στην Σουηδία με τη νέα νομοθεσία που ισχύει από τον Ιανουάριο του Τρέχοντο. Άλλα σημαντικά στοιχεία είναι τα θέματα της εμπιστευτικότητας, της ταυτότητας του ε, καταγγέλλοντος και η προστασία από ε, αντίπεινα. Αυτά είναι πολύ σημαντικά στοιχεία και θα πρέπει να αναφέρονται ρητά στις καλές πρακτικές και στην νομοθεσία. Δεν παρέχουν όλα τα κράτη-μέλη ε, ρήτρε για την ε, ε, προστασία της ταυτότητας του καταγγέλλοντος. Επίσης, ο καταγγέλλον έχει πρόσβαση σε ανεξάρτητες αρχές για την παροχή ας πούμε, Υπάρχουν κάποιοι φορείς, κάποια κρατημέλη που προσφέρουν στους καταγγέλλοντες συμβολή, βοήθεια, πού πρέπει να απευθυνθούν, ποιε είναι οι νομικέ προστασίε που μπορεί να έχουν, τι αντίπεινα μπορεί να αντιμετωπίσουν κλπ. Και επίση η υποπτία, η αναθεώρηση και η αξιολόγηση. Και εδώ φτάνω στο τελευταίο μου σημείο για την εφαρμογή των νόμων, έστω και αν είναι πλήρε. Στην πράξη βλέπουμε ότι δεν εφαρμόζονται πάντα είτε γιατί δεν είναι γνωστοί στον ιδιωτικό τομέα. Πρόσφατα μια μελέτη του ΩΣΑ ε, δείχνει ότι 83% περίπου δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει δυνατότητα να κάνουν την καταγγελία του εσωτερικά ή επειδή η νομοθεσία δεν εφαρμόζεται γενικώ στην πράξη. Οπότε η αξιολόγηση και η αναθεώρηση θα πρέπει να είναι σημαντικέ, έτσι ώστε να απομακρυνθούμε από μια απλώ καλή νομοθεσία στα χαρτιά και να περάσουμε σε μια καλή νομοθεσία που όντω θα βοηθάει του καταγγέλλοντες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Αμπάτση. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας, ιδιαίτερα για το παράδειγμα για τις βέλτιστες πρακτικές της Ιρλανδίας. Θα δώσω το λόγο τώρα στην Σαρλότα Γκράς. Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας σήμερα για να μεταφέρω τις απόψεις των επιχειρήσεων Εκπροσωπώ την εταιρεία Valorec, γαλλική εταιρεία δραστήρια στον τομέα των σωλήνων από χάλιβα και επίσης την Ένωση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων που αποτελείται από 8 εκατομμύρια εργαζομένων στον κόσμο και 100 ε, δις κύκλο εργασιών. Να πω ότι καταρχάς είμαστε υπέρ της δημιουργίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενός διατομεακού α, μέσου. Όπως είπαμε σήμερα έχουμε διαφορετικά συστήματα στα κράτη-μέλη και είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις ευρωπαϊκού επίπεδου που έχουν μισθωτού σε διάφορες χώρες της Ένωσης να κάνουν ρυθμίσεις στο εσωτερικό τους για την προστασία των καταγγελόντων και να μπορούν να είναι συμβατές οι ρυθμίσεις αυτές με τις διαφορετικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Υπάρχει επίσης μερικές φορές και το θέμα της αντίθεσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τις Ηνωμένε Πολιτείες σαν παράδειγμα αν το σύστημα προστασίας των καταγγελόντων δεν είναι συμβατό με τις αμερικανικές διατάξεις. Πάντως είναι σημαντικό το σύστημα προστασίας <clears throat> για να ξεκινήσει να είναι ένα σύστημα το οποίο θα πρέπει να καθοριστεί με πολύ συγκεκριμένο τρόπο έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα. τώρα για τον ορισμό ε, του καταγγέλλοντος. Ε, ε, εγώ παραπέμπω στο νόμο ΣΑΠΑ 2, έγινε δεκτό στη Γαλλία το Δεκέμβριο του 2016, δημιουργεί ένα καθεστώς διατομεακό όπως είπα και με λίγες επιφυλάξεις αποτελεί, θα έλεγα ή θα αποτελούσε έστω μια καλή βάση και για ένα κοινοτικό μέσο. Τώρα για τον ορισμό μου φαίνεται σημαντικό ο καταγγέλων να βρίσκεται σε σχέση εργασίας με την επιχείρηση. Θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει οικονομικό συμφέρον, δεν θα πρέπει να υπάρχει αμοιβή για την καταγγελία, γιατί αλλιώς θα μπορούσαμε να έχουμε στρεβλώσεις του συστήματος. Ε, σύμφωνα με το γαλλικό νόμο, ο καταγγέλων θα πρέπει να είναι καλής πίστεως και να γνωρίζει ακριβώς τα τεκτενόμενα και να μην βασίζει τις καταγγελίες του σε φήμες. Για το πεδίο της προειδοποίησης θα πρέπει να είναι διατομεακό, αλλά να περιορίζεται και σε θέματα σοβαρών παραβιάσεων του νόμου, είτε στον τομέα του ανταγωνισμού, των περιβάλλων, τις εργασιακές σχέσεις κτλ. Σχετικά τώρα με τους διάβλους καταγγελίας, έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα, θα έλεγα, βαθμιαίο σύστημα, το οποίο θα δίνει την δυνατότητα καταρχάς να ενημερώνει ο καταγγέλων την ίδια την επιχείρηση, είναι ένα σύστημα το οποίο υπάρχει στη Γαλλία, επιβάλλει συγκεκριμένα μέτρα στις επιχειρήσεις ε, σχετικά ε, με την παραδοχή αποδοχή μάλλον της καταγγελίας, καταγραφή της αποδοχής ε, και μόνο σε περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση δεν κάνει κάτι, τότε οι καταγγέλλοντες μπορούν να προσφύγουν στις τοπικές αρχές, ε, ε, στις εργασιακές αρχές ή στην δικαιοσύνη αλλά θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα όμως να έχουν ε, και ε, πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης. Τώρα, σχετικά ε, με τις διαδικασίες και τους διάβλους καταγγελίας, υπάρχουν επιχειρήσεις διαφορετικής τυπολογίας, διαφορετικού μεγέθους και με διαφορετικά μέσα. Είναι σημαντικό πλαισιώνοντας αυτές τις επιχειρήσεις με κοινέ υποχρεώσεις να τους δίνουμε την δυνατότητα να δημιουργούν διαδικασίες προσαρμοσμένες στην επιχείρηση έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματικές ε, στο εσωτερικό τους και σε σχέση με τα μέσα και σε σχέση με την επικοινωνία και την ενημέρωση των εργαζομένων. Ένα τελευταίο σημείο το οποίο θα ήθελα να θέσω Ζητάμε από τις επιχειρήσεις σήμερα να δημιουργούν όπως είπα τα συστήματα τα οποία θα επιτρέπουν να γίνονται εσωτερικές έρευνες. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να οδηγήσει και σε κυρώσεις εσωτερικές, να οδηγήσει και σε προσφυγές σε δικαστικά συστήματα. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει μόνο στη Γαλλία. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι ικανές πάντως ε, να προωθήσουν τέτοιου είδους έρευνες στο εσωτερικό της επιχείρησης. Ευχαριστώ κύριε Κρά. Σας ευχαριστώ και για τις γραπτές παρατηρήσεις που μας έχετε στείλει ε, που θα επιτρέψουν και σε όλους τους συναδέρφους να ε, διαβάσουν αυτά που είπατε. Δίνω τώρα το λόγο στην Κάθη James, που προέρχεται από μη κυβερνητική οργάνωση που ασχολείται με ε, τις δημόσιες υπηρεσίες. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ την Επιτροπή σας που με κάλεσε ε, εδώ να μιλήσω σήμερα. Μιλώ για τον οργανισμό Public ε, Concerns at Work, διότι ασχολούμαστε με το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ανθρώπους να καταγγείλουν παρατυπίες στον χώρο εργασίας. Δημιουργηθήκαμε πριν περίπου 25 χρόνια. Μετά από μεγάλα ε, επιχειρηματικά σκάνδαλα, την ε, κατάρρευση μεγάλων τραπεζών, ε, το καταστροφές σε πλοία, διαπιστώσαμε ότι σε όλες τις περιπτώσεις το προσωπικό γνώριζε. Άνθρωποι που εργάζονταν εκεί το ήξεραν, αλλά είτε φοβούνταν ε, να το καταγγείλουν ε, λόγω της κουλτούρας ε, που υπήρχε στον χώρο εργασίας ή είχαν διαμαρτυρηθεί και κανείς δεν έκανε τίποτα. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι θα είναι χρήσιμο να παρέχετε βοήθεια σε πρόσωπα δεν... Το θέμα είναι ότι ο εργαζόμενος δεν ξέρει σε ποιον να υποβάλει αναφορά, πώς να το κάνει, πότε κλπ. Παρέχουμε συμβουλές λοιπόν ε, σε άτομα και έχουμε παράσχει σε 25.000 άτομα συμβουλές ε, και έχουμε απαντήσει σε 46.000 αιτήματα για σύμβουλες. Κάνουμε διάκριση ανάμεσα στα θέματα δημοσίου συμφέροντος ε, και τα υπόλοιπα. Στόχος μας είναι οι πληροφορίες να μεταφερθούν σε κάποιον που να μπορεί να επαναρθώσει την κατάσταση και αν όχι ε, να γίνει κάτι για αυτό. Για παράδειγμα, ε, η πώληση πώληση τροφίμων ακατάλληλων σε σούπερ μάρκετ, ε, λήψη δειγμάτων αίματος ε, για ε, τεστ για AIDS χωρίς τη συγκατάθεση του εργαζομένου, να δοκιμάζονται οι αντιδράσεις φοιτητών σε ζωντανό ασθενή. Βλέπουμε λοιπόν πώς οι διάφορες επιχειρήσεις προσπαθούν να ξεφύγουν και βλέπουμε και περιπτώσεις όπου πράγματι εισακούονται ε, όπου μάλλον ε, ακούνε τις ανησυχίες ε, των εργαζομένων, αλλά τα τρία τέταρτα των ανθρώπων που έρχονται σε εμά λένε ότι δεν έχει γίνει τίποτα για να διορθωθεί η κατάσταση. Παρέχουμε συμβουλές, υπάρχει και νομοθεσία στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 1998, αλλά η δικαστική ε, οδόση είναι μόνο μέρος των συμβουλών που δίνουμε. Είναι σημαντικό σε περίπτωση που δεν πάνε καλά τα πράγματα, να έχει κανεί το δικαίωμα αυτό, ε, αλλά ε, προσπαθούμε να παρέχουμε πρακτικές συμβουλές. Συνεργαζόμαστε και με διάφορους οργανισμούς και προσπαθούμε να τους κάνουμε να σκεφτούν τις ε, δομές διαχείρισης ε, και ανάλυσης κινδύνου. Θα πρέπει να θεωρεί κανείς δώρο ε, έναν εργαζόμενο που καταγγέλει παρατυπίες εντός του οργανισμού του. Και θα πρέπει να προστατεύει τους ανθρώπους αυτούς ο οργανισμός καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Το να προσπαθήσουμε λοιπόν να δείξουμε στις επιχειρήσεις και σε άλλους οργανισμούς πώς έχουν τα πράγματα αποτελεί ε, επίσης μέρος της δουλειάς μας. Είχαμε πρόσφατα σκάνδαλα σε σχεδόν όλους τους τομείς, σε τράπεζες, στην υγεία, είχαμε το σκάνδαλο της Volkswagen, ε, είχαμε το σκάνδαλο με το κρέας αλόγου. Φαίνεται σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα τελικά. Η δουλειά που κάνουμε λοιπόν είναι εξίσου σημαντική τώρα όσο ήταν πριν 25 χρόνια όταν ε, ιδρύθηκε ο οργανισμός μας. Τώρα νομίζω υπάρχει περισσότερο ενδιαφέρον στους καταγγέλλοντες, για τους καταγγέλλοντες παρατυπίες. Άλλωστε ζούμε στην εποχή του διαδικτύου, έχουμε τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Όλα αυτά καθιστούν πολύ σημαντικό ε, ε, η προστασία των καταγγελόντων παρατυπίες ε, να γίνεται και διασύνοριακά. Θα πρέπει να μπορούμε να ε, λέμε την αλήθεια απέναντι στους ηθήνοντες. Πρέπει όμως να γίνει δουλειά ευαισθητοποίησης του κοινού πάνω στο θέμα αυτό. Αυτό λείπει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, η κυβέρνησή μας ε, θέσπισε τον νόμο, δεν έκανε όμως ε, τίποτα για να τον προωθήσει. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της ευαισθητοποίησης του κοινού. Μόνο το 26% των εργαζομένων στο Ηνωμένο Βασίλειο γνωρίζουν ότι υπάρχει νόμος που τους προστατεύει. Φροντίστε λοιπόν ε, να ευαισθητοποιηθεί και το κοινό απέναντι στα προβλήματα αυτά. Επίσης, ο ε, ε, κατά κέλων παρατυπίες δεν είναι σαν αυτούς ε, για τους οποίους διαβάζετε σε εφημερίδες. Ε, λέει κάτι μία-δύο φορές, ε, αλλά μετά εγκαταλείπει τον αγώνα και παρετείται από την προσπάθεια. Ανησυχητικό είναι ότι την τρίτη φορά που αποφασίζει κανείς να καταγγείλει κάτι, ο οργανισμός θα ακούσει τι έχει να πει. Στο Ηνωμένο Βασίλειο Γίνεται προσπάθεια στον τομέα της υγείας, ε, για παράδειγμα, να κλείσει το κενό αυτό. Αλλά το πρόβλημα του νόμου στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ότι προβλέπει αποζημίωση προς το άτομο, αλλά σημαίνει ότι το άτομο θα πρέπει να ασκήσει το δικαίωμα αυτό. Επίσης ε, δεν ε, απαιτείται τίποτα από τους ρυθμιστές από τη στιγμή που θα λάβουν ε, παρατηρήσεις ή πληροφορίες για αμυρατυπία. Πρέπει λοιπόν αφενός να οριστεί τι είναι ο καταγγελόν παρατυπίες, δεύτερον να διαπιστωθεί τι μπορεί να γίνει στην περίπτωση που υπάρχει ένα περιστατικό. Το βάρος απόδειξης θα πρέπει να έχει όσο γίνεται πιο χαμηλό κατόφλι, το βάρος θα πρέπει να το φέρει ο εργοδότης. Και είναι πολύ σημαντικό να παρέχονται συμβουλέ. Δεν ξυπνάει κανεί το πρωί και λέει ότι Α, σήμερα θα γίνω καταγγέλων παρατυπίε. Είναι κάτι που διαπιστώνουν ότι γίνεται επανειλημμένα στον χώρο εργασία του και πρέπει να βοηθήσουμε του ανθρώπου αυτού. Σα ευχαριστώ πολύ, κυρία Τζέιμ. Η μη κυβερνητική οργάνωσή σα ε, είναι μια από τις σημαντικές οργανώσεις ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Διαβάζω εδώ ότι έχετε πάνω από 2.000 υποθέσεις το χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην καθηγήτρια Φρεντερίκ Πέρο. Παρακαλώ. Merci beaucoup. Merci beaucoup de... Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή που θα δείξετε. Θα ήθελα να αναφερθώ στο πρόβλημα στα πλαίσια μιας νομικής ρύθμισης που να επιτρέπει την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να διευκρινίσω ότι η έννοια του καταγγέλλοντος εξελίσσεται και στα κράτη-μέλη και στο εσωτερικό του Συμβουλίου της Ευρώπης έτσι ώστε να θεωρηθεί ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο παίζει δημοκρατικό ρόλο και καταγγέλει ε, τις δυσλειτουργίες ε, γενικότερα τις διοικητικές δομές των διοικητικών δομών. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σαφές ότι το πρόβλημα σήμερα είναι ένα πρόβλημα διαφοροποίησης των εθνικών αντιμετωπίσεων, κάτι το οποίο δημιουργεί, αν θέλετε, πρόβλημα στην σύλληψη ε, των διαφορετικών μορφών προστασίας του καταγγέλλοντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια πολύ διασπασμένη αντίληψη για το πρόβλημα. Υπάρχει μια κάποια προστασία η οποία είναι όμως πολύ ε, ε, επιμερισμένη και τομεακή και θα πρέπει να υπάρξει μια προσπάθεια έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το επίπεδο προστασίας και να καλυφθούν τα νομικά κενά. Νομίζω ότι το δεύτερο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι η δημιουργία κάποιων επίσημων διαδικασιών σύμφωνα με την ομολογία του Δικαστηρίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει να υπάρξει μια οριζόντια αντιμετώπιση λοιπόν. Αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προστατευτεί ταυτόχρονα η δημοκρατία, η ελευθερία έκφρασης, κάτι το οποίο σε νομικό επίπεδο με βάση τις συνθήκες είναι ίσως και ανέφικτο. Μια οριζόντια λοιπόν αντιμετώπιση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί επί τη βάση του 114 των συνθήκων που διέπει την εσωτερική αγορά και που έχει το πλεονέκτημα στον τομέα της λήψης των αποφάσεων να παρουσιάζει πλεονεκτήματα ε, μεταξύ των οποίων και την ενισχυμένη πλειοψηφία στις λήψεις αποφάσεων του Συμβουλίου. Κάτι θα μας επέτρεπε τέτοιο να λύσουμε τις διαφορές ανάμεσα στις εθνικές μορφές αντιμετώπισης. Το πρόβλημα του 114 είναι ότι πρέπει να αποδείξει ότι ο ορισμός του καταγγέλλοντα είναι αναγκαίος για να λειτουργήσει η εσωτερική αγορά. Συγγνώμη που αρχίζω και μπερδεύω λίγο τα άρθρα της συνθήκης να αναφερθώ στο 352 την ρήτρα ευελιξίας δηλαδή που επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλαμβάνει δράση ακόμα και όταν δεν έχει το σύνολο των εξουσιών στην διάθεσή της και πρέπει να παραμείνει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της. Το 352 ως έχει δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον του διότι θα πρέπει να ισχύσει σε διάφορες πολιτικές σε συνδυασμό με το 114, το οποίο θα επιτρέψει να διευρύνουμε τις δράσεις που μπορούμε να αναλάβουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία των καταγγελόντων. Αυτή η συνδυαστική αντίληψη είναι ενδιαφέρουσα γιατί θα επιτρέψει μια ευρεία μορφή ορισμού του καταγγέλλοντα και των δικαιωμάτων του καταγγέλλοντα. Ε, σας θυμίζω ότι στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης υπάρχει το δικαίωμα στην εμπιστευτικότητα, στην επαρκή αντιμετώπιση ε, ε, του προβλήματος από πλευράς της επιχείρησης ή των δημοσίων αρχών και το δικαίωμα του καταγγέλλοντα να είναι ενήμερος για τη συνέχεια που δίδεται στην ενέργεια την οποία κάνει όπως επίσης και να υπάρχει ένα πλαίσιο μέτρων που να απαγορεύει τις κυρώσεις εις βάρος του καταγγέλλοντα. Λοιπόν, το 114 με το 352 μπορούν να προασπίσουν την αντίληψη που λέγει ότι η προστασία του καταγγέλλοντα είναι τμήμα της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης των επιχειρήσεων. Και αυτό είναι προϋπόθεση έτσι ώστε οι επιχειρήσεις αυτές να εποφελούνται από την εσωτερική αγορά στα πλαίσια μιας λογικής την οποία συναντάμε ε, και στο εδάφιο 8 της οδηγίας ε, για την εμπιστευτικότητα και το απόρριτο των εμπορικών συναλλαγών. Μπορεί να υπάρχει επίσης και μια υπερτοπική αντιμετώπιση γιατί κάποιες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όπως γαλλικές επιχειρήσεις έχουν να καλύψουν κάποιες απαιτήσεις για την προστασία των καταγγελόντων που μπορεί να είναι είτε διεθνής είτε η αμερικανική λογική αν θέλετε που έχει επιπτώσεις και στις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Προφανώς το πρόβλημα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει στην παρούσα φάση η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η έννοια της επικουρικότητας, η αρχή της επικουρικότητας όχι μόνο σε νομικό επίπεδο, αλλά είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη επίσης τη σύνδεση με τις εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις, από τις οποίες θα έλεγα παίρνουν στοιχεία και οι διεθνείς προσπάθειες κάλυψης. Ε, εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε να είναι ένα βήμα δικαίου, μια έδρα δικαίου αν θέλετε, που θα επιτρέψει στις ε, χώρες να καλύψουν το νομικό κενό. Τώρα για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αποζημίωσης είναι κάτι που θα δημιουργήσει πρόβλημα στην αρχή της επικουρικότητας. Το πρόβλημα που μπορεί να δημιουργήσει λοιπόν είναι ότι θα υποχρεωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει μέρος, αν θέλετε, ε, με τη μία ή άλλη πλευρά, κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο και γι' αυτό πιστεύω ότι δεν είναι διαπραγματεύσιμο το θέμα της αποζημίωσης μέσω κοινοτικού ταμείου. Θα πρέπει να μην αγνοήσουμε και τις υπόλοιπες αντιλήψεις όπως την διακανονιστική, νομική, έχει κάποια θετικά στοιχεία, απαιτούνται κατευθυντήριες γραμμές στην Ένωση, για να προασπιστεί η ιδέα και της διακυβέρνησης των επιχειρήσεων αλλά και της ε, ε, θα έλεγα δημοκρατικής νομιμότητας, ε, νομιμοποίησης συγγνώμη, των μέτρων προστασίας. Σας ευχαριστώ κυρία Μπερό. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Χίτλη είναι υπεύθυνη για θέματα εσωτερικής στρατηγικής και κανόνων στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Θα μας πείτε πώς αυτό επηρεάζει και λειτουργεί στις ευρωπαϊκές, στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που καλέσατε το γραφείο του Διαμεσολαβητή για να σας ενημερώσει για τι κάνουμε εμείς στην τομέα αυτό. Θέλω θέλω να σας μιλήσω για, την, ε, για το ρόλο και την εντολή. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγει τον ε, Ευρωπαϊκό Δημοσιολαβητή και το 2013 εξέλεξε την Εμιλία Ράιλι. Διερευνούμε την κακοδιαχείριση στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τους φορείς, τις υπηρεσίες, και επί τη βάση των καταγγελιών που έρχονται από πολίτες ή από μέσω ερευνών ιδίως πρωτοβουλίας. Οι ομάδε μα, οι διερευνητικέ ομάδε, έχουν εξουσία να ε, εξεργάζονται όλα τα έγγραφα που έχουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και να ζητούν την κατάθεση Ευρωπαίων ε, υπαλλήλων των θεσμικών οργάνων. Ε, τακτικά, σε τακτικά διαστήματα ελέγχουμε τα έγγραφα αυτά και έχουμε καλή συνεργασία με τα θεσμικά όργανα σε ό,τι αφορά την εξαγωγή των ελέγχων, των ερευνών και τη διευκόλυνση της δουλειάς μας σε καθημερινή βάση. Πάνω από 90% των ερευνών μας βασίζονται σε καταγγελίες και τα μέλη του κοινοβουλίου σας μπορούν βεβαίως να στείλουν καταγγελία στην, ε, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή αν θέλουν ας πούμε, πρόσβαση σε ε, ευρωπαϊκά έγγραφα. Τα θεσμικά όργανα βεβαίως ε, συμμορφώνονται περίπου στο 85-90% με τις συστάσεις του Διαμεσολαβητού. Γενικώ λοιπόν αυτά για τη δουλειά μας. Τώρα για το θέμα που θέλουμε να συζητήσουμε σήμερα. Όντω θα σα μιλήσω και εγώ για την ε, στρατηγική έρευνα του Διαμεσολαβητή, αλλά και για τη δική μα εμπειρία ω ε, υπηρεσία σε ό,τι αφορά την ε, προστασία των καταγγελόντων. Και θα σα δείξω βεβαίω τη δική μα την εμπειρία σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των καταγγελιών από καταγγελίε. Και τι είδου καταγγελίε έρχονται στον διαμεσολαβητή. Μία από τις βασικές στρατηγικές έρευνες ε, της ε, κυρίας Οράιλη ήταν ε, ακριβώς για το θέμα αυτό των καταγγελιών. Και υπήρχε καταρχάς το, η πρώτη έκθεση για την αντιμετώπιση της διαφθοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί αναφέρεται ότι οι, καταγγελίες, οι καταγγέλλοντες αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες για την αναφορά τέτοιων κακών διαχειρήσεων λόγω ακριβώς της, του φόβου αντιπίνων. Και βεβαίω πρέπει να δημιουργηθεί μια κουλτούρα ε, ακαιρεότητας εντός των θεσμικών οργάνων, να αυξηθεί ναι, η ναι. ευαισθητοποίηση και να δημιουργηθούν μηχανισμοί που θα δώσουν εμπιστοσύνη, ε, έτσι ώστε να μπορούν οι καταγγέλλοντε να κάνουν την καταγγελία τους. Αυτό λοιπόν θεώρησε ότι είναι πολύ σημαντικό η α, διαμεσολαβήτρια και γι' αυτό το προώθησε. Ε, ξεκίνησε λοιπόν ο σχετικό κανονισμό, ήδη από τον... υιοθετήθηκε το 2014 και στο άρθρο 22C ε, αναφέρονται οι ιστορικοί κανόνες ε, που καλύπτονται η ανάγκη για παροχή πληροφοριών στους ε, υπαλλήλου, για τη διαχείριση θεμάτων που καταγγέλλονται. Η προστασία επίσης των νόμιμων συμφερόντων των συγκεκριμένων αυτών υπαλλήλων και τη ιδιωτικότητά του και η διαδικασία για τη διαχείριση καταγγελιών από υπαλλήλου ε, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίου ε, τους, τους μεταχειρίστηκαν. Αυτές οι διατάξεις νομίζω ε, αποδεικνύονται και από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει και διαχειρίζεται η διαμεσολαβήτρια της καταγγελίας αυτέ. Τα περισσότερα παράπονα έρχονται από άτομα που δεν, λένε ότι δεν τους πήραν στα σοβαρά όταν έκαναν την καταγγελία τους, ότι η ιεραρχία τους δεν ακολούθησε τις, ε, τα όσα είπαν, ότι δεν είχαν καμία ενημέρωση μετά για το αν ελήφθη κάποια δράση, κάποιο μέτρο. Είχαν λοιπόν πολύ λίγη ανταπόκριση για το κατά πόσο ήταν όντως ε, σωστή η καταγγελία που έκαναν. Και συμφωνώ με αυτό που είπε και η ε, συνάδελφος γιατί όντως ε, δείχνει ότι πραγματικά συμβαίνει αυτό και στα κρατη τουλάχιστον στο Ηνωμένο Βασίλειο συμβαίνει σίγουρα. Και τέλος, οι καταγγέλλοντες έρχονται στο δικό μας το γραφείο όταν αντιμετωπίζουν αντίπεινα. Με αυτές λοιπόν τι ε, διατάξεις η δημοσιογραφική ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την υπηρεσία την αναλάβει τον ηγετικό ρόλο έτσι ώστε να εκπονήσει εσωτερικού κανόνε. Και βεβαίω βοηθηθήκαμε από τα στοιχεία που βλέπετε στη διαφάνεια, ότι ε, η, μια αποτελεσματική πολιτική θα πρέπει να ε, αποτρέπει και να εντοπίζει την ε, κακοδιαχείριση πριν συμβεί, να δείχνει ότι η ανώτατη ιεραρχία θέλει να ακούσει τι ανησυχίε που έχουν οι υπάλληλοι ήδη από την αρχή και να απαντήσει α, αναλόγως. Θα πρέπει να δείχνει στο προσωπικό πώς να θίξει ένα τέτοιο είδος πρόβλημα έτσι ώστε να είναι σαφή η διαδικασία. Θα πρέπει να εξασφαλίζει, να ε, επιβεβαιώνει στο, στο προσωπικό ότι θα προστατευτεί εάν υπάρξουν καταγγελίε, ότι βεβαίω θα πρέπει να υπάρχουν ε, ε, συγκεκριμένε πληροφορίε για του τους υπόλοιπου τρόπου η υποβολή μια καταγγελία, όλα α πούμε οι άλλε υπηρεσίε, και να μειώνεται το, ο κίνδυνο για την δημοσίευση αυτών των πληροφοριών. Μιλάμε βεβαίω τώρα για, τους, για, την, όλη την ε, ιεραρχία, από τους ε, πιο υψηλά ιστάμενους μέχρι τους ε, κατώτερους υπαλλήλους, Όλο το, όλο το προσωπικό λοιπόν πρέπει να γνωρίζει τους κανόνες, να ε, ξέρει πώς ακριβώς λειτουργούν και γι' αυτό η, ε, η έρθει σε επαφή με την ε, Επιτροπή του σχετικού, την Επιτροπή που ασχολείται με τα θέματα αυτά από την πλευρά του προσωπικού και θεωρήσαμε ότι τα, οι κανόνες αυτοί θα έπρεπε να μπουν και σε μια δημόσια διαβούλευση και η ε, οργάνωση της κάθε επίσης έστειλε τις απόψεις της καθώς και άλλες και έτσι ολοκληρώσαμε μετά από αυτή τη διαβούλευση την, α, τους κανόνες και μετά ξαναπήγαμε στην Επιτροπή του Προσωπικού για να δούμε αν συμφωνούν με τη θέσπιση αυτών των κανόνων. Δεν θα σας πω τώρα τις λεπτομέρειε των κανόνων, υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας και έχω απαντήσει ήδη στις ερωτήσεις που έβαλε η Επιτροπή σας. Ε, έχουμε, έχουμε όμως τους ορισμούς, έχουμε τη διαδικασία, πώς διεξάγεται, έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία όπως το ότι ο καταγγέλων προστατεύεται, ότι είναι σημαντικό να μην υπάρχει κατάχρηση της διαδικασίας, τα δικαιώματα του ατόμου που εμπλέκονται και όλα αυτά τα στοιχεία. Αφού λοιπόν κάναμε τους δικούς μας ε, κανόνες και καθαρίσαμε τα του οίκου μας, ε, η διαμεσολαβήτρια ξεκίνησε να ρωτά τι κάνουν τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Μόνο δύο από τα εννέα που μελετήσαμε είχαν κανόνες συγκεκριμένους η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο συγκεκριμένα. Λίγο μετά την ολοκλήρωση της ερευνάς από τη Διαμεσολαβήτρια και τα εννέα θεσμικά όργανα είχαν εισαγάγει τέτοιους κανόνες συμπεριλαμβανομένου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οπότε, εμείς δεν είδαμε την ουσία των ε, κανόνων του κάθε θεσμικού οργάνου ξεχωριστά, αλλά γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό που είμαστε σήμερα εδώ, γιατί έτσι μπορούμε να κάνουμε μάλλον το ε, επόμενο βήμα από την πλευρά του γραφείου του, του να ανταλλάξουμε τις εμπειρίε μας και να δούμε πώς εφαρμόζονται τελικά οι κανόνες. Και βεβαίως, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μας καλέσατε εδώ για να μπορέσουμε όλα αυτά να τα συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Χεκή. Λάβαμε μια πολύ καλή επισκόπηση. Από την καθηγήτρια Απάτση είχαμε μια γενική επισκόπηση. Από την κυρία Κράς από τη Γαλλία λάβαμε αποτελέσματα, παραδείγματα. Από την κυρία Τσέις για το Ηνωμένο Βασίλειο, από την ε, κυρία Περό μάθαμε τις πρακτικές ε, εντός του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επισκόπηση. Θα, ακούσουμε, θα περάσουμε τώρα στις ερωτήσεις ε, και παραδίδω την Προεδρία ε, στον συνάδελφο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε τα όσα είπαν οι εμπειρογνώμονες. Ε, ήρθε τώρα η σειρά των Ευρωβουλευτών να πάρουν το λόγο. Η κυρία Βιρζινή Ροζιέρ πρώτη για πέντε λεπτά το πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να εκμεταλλευτώ με τον καλύτερο τρόπο τον χρόνο που μου δίνεται και να θέσω ερωτήσεις προς τις ομιλητριές μας. Προς την κυρία Αμπάζη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία στα κράτη-μέλη. Αλλά θα μπορούσα να απευθύνω αυτή την ερώτηση και προς την κυρία Τζέιμς που έχει πρακτική εμπειρία παρέχοντας βοήθεια στους καταγγέλλοντες παρατυπίες ο καλύτερος τρόπος να περιγράψουμε την κατάσταση. Ε, δείχνει ότι θα πρέπει να βρούμε έναν ορισμό και θα πρέπει αυτός ο ορισμός να βασιστεί στο είδος της καταγγελίας, στο είδος της απάτης, αν πρόκειται για χρηματοοικονομική απάτη ή θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στο στόχο, στο δημόσιο συμφέρον για παράδειγμα και να έχουμε όσο γίνεται πιο ευρεία προσέγγιση και να καλύψουμε όσο γίνεται περισσότερες περιπτώσεις. Πρέπει να βρούμε έναν όσο γίνεται πιο σαφή ορισμό. και να μπορούμε να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα σε κάποιον καταγγέλλοντα παρατυπίες για ηθικούς λόγους και σε κάποιον που απλά διοχετεύει πληροφορίες που δεν θα έπρεπε. Και υπάρχει και το θέμα της καλής πίστης. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας και μάλιστα όλων των ομιλητριών για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι χρειάζεται το θέμα αυτό όχι απαραίτητα για τον ορισμό των καταγγελόντων, αλλά για να καλύψουμε περιπτώσεις όπου η καταγγελία έγινε καλή την πίστη, αλλά όπου δεν ε, έχουν αποδειχθεί οι καταγγελίες μπορεί κάποιος να καταγγείλει παρατυπίες, ε, να μην ε, βρεθούν στοιχεία, να μην αποδεχτεί ότι πράγματι υπάρχουν παρατυπίες, αλλά αυτή η καταγγελία να έχει γίνει καλή τυπίστη και θα πρέπει να παρέχεται προστασία στην περίπτωση αυτή. Προς την κυρία Κράς. Υποβάλλατε συστάσεις ε, σχετικά με το τι θα πρέπει να γίνει. τι κάνουν οι διεπιχειρήσεις, τι όχι και πόσο μπορούμε να θεσπίσουμε κανόνες ώστε αυτό να γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αν υπάρχει κάποιος που είναι διατεθειμένος να μεταφέρει πληροφορίες, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τις πληροφορίες αυτές για να βελτιώσουμε την εσωτερική λειτουργία της επιχείρησης. δεν θα είχαμε κάνει πρόσφατα όλες ε, τις συζητήσεις που είχαμε τα τελευταία χρόνια, εάν είχαμε θεωρήσει ότι μπορούμε να καλύψουμε μόνο τις περιπτώσεις που ρητά αναφέρονται στο δίκαιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποια ευελιξία. Τι προσέγγιση θα πρέπει να επιλέξουμε. Είναι αλήθεια ότι εάν περιορίσουμε το πεδίο εφαρμογής ε, στην εσωτερική αγορά μπορεί να είναι πιο εύκολα τα πράγματα για μας, αλλά μήπως ε, θα πρέπει να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής. Ε, θα είναι βέβαια αυτό κάτι πιο πολύπλοκο, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε όλες τις δυνατότητες. Και τέλος, προς την εκπρόσωπο του γραφείου της διαμεσολαβήτριας. Αν καταφέρουμε να σημειώσουμε πρόοδο και καταφέρουμε να έχουμε προστασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ε, σήμερα η εντολή της διαμεσολαβήτριας ε, περιορίζεται στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θα μπορούσαμε όμως να διευρύνουμε την, το πεδίο, την εντολή σας ώστε να καλύπτει και τους οργανισμούς που λαμβάνουν αναφορές από κατακέλλοντες. Ε, πιστεύετε ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια πιθανότητα να διευρύνουμε τις εξουσίες της διαμεσολαβήτριας. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Ελπίζω να τήρησα το χρόνο μου. Δεν ε, ε, είχα καταλάβει καλά. Με ενημερώνω ότι πέντε λεπτά πρέπει να είναι η ερώτηση μαζί με την απάντηση. Αλλά θα ακούσουμε και τους άλλους δύο συνεισηγητές και κατόπιν θα δώσουμε το λόγο στις εμπειρογνώμονες για να απαντήσουν. Ο κύριος Κόφοντ, παρακαλώ ε, να λάβετε υπόψη σας την πίεση χρόνου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Άλλωστε έχουμε συνηθίσει να εργαζόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Θα είναι σύντομες οι ερωτήσεις μου για να υπάρχει χρόνος να ακούσουμε τις απαντήσεις. Καταρχάς ε, θα ήθελα να πω ότι είμαστε μέλη της Επιτροπής ΠΑΝΑ μόνο και μόνο επειδή υπάρχουν άνθρωποι απατεώνες, έχουμε παραδείγματα κακοδιαχείρισης κλπ. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το να συζητάμε το θέμα των καταγγελόντων παρατυπίες. Και βλέπετε στην Ευρώπη γίνεται χαμός. Ε, υπάρχει λοιπόν πολύ ε, περιθώριο δράσης για μας. Η ερώτησή μου, έχετε παραδείγματα των πρακτικών αναχώρα. Έχετε αναφέρει κάποιες στις γραπτές σας απαντήσεις και θα ήθελα επίσης να ακούσω τις χείριστες πρακτικές και επίσης σε επίπεδο επιχειρήσεων θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Στην περίπτωση των Lux Leaks, ε, ο καταγγέλων και ο δημοσιογράφος καταδικάστηκαν, ε, διώθηκαν δικαστικά, ενώ η επιχείρηση ε, υπέστη πολύ περιορισμένες κυρώσεις. Και επίσης κυρία Περό, ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε για τη νομική βάση για μια οριζόντια προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορείτε να το αναπτύξετε αυτό. Πώς μπορούμε να έχουμε ε, πλαίσιο ευρωπαϊκού επίπεδου για την προστασία των κατακελώντων και πώς μπορούμε να απαιτήσουμε από τα κράτη-μέλη να διασφαλίζουν καλύτερη προστασία σε εθνικό επίπεδο. Τι δυνατότητες και τι περιορισμούς βλέπετε όσον αφορά το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ιεζέκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα. Εάν ε, σκεφτούμε τις αποκαλύψεις ε, για τα έγγραφα του Παναμά, ε, ένα από τα σημαντικότερα θέματα είναι η ανωνυμία κατά την καταγγελία παρατυπιών. Ερώτηση προς την καθηγήτρια Απάζη όσον αφορά την αποζημίωση. Είτε είναι ψυχολογική υποστήριξη είτε οικονομική βοήθεια. Τι διαφορές υπάρχουν ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Προς την κυρία James. γνωρίζουν ε, οι άνθρωποι πώς μπορούν να καταγγείλουν κάποια παρατυπία, πώς μπορούμε να διευκολύνουμε τις καταγγελίες. Προς την κυρία Περό, όσον αφορά το βάρος απόδειξης ανάμεσα στον καταγγέλλοντα και στον εργοδότη. Και προς την κυρία Χίκη, τα θεσμικά όργανα υιοθέτησαν και αναβάθμισαν τους εσωτερικούς κανόνες. Πώς εφαρμόζονται αυτοί οι κανόνες. Και η κυρία Κράς ήδη αναφέρθηκε στον εσωτερικό μηχανισμό. Δεν έχω ερωτήσει λοιπόν σχετικά με αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε τώρα παρακαλώ να περάσουμε στις απαντήσεις. Παρακαλώ. Με όποια σειρά θέλετε. Να δώσουμε πρώτο το λόγο στην κυρία James. Ευχαριστώ. Πολύ σημαντικά τα όσα είπατε για τους ορισμούς ε, εντός των ιστορικών κανονισμών που έχουν αντιμετωπίσει τέτοια θέματα εντός της ε, νομοθεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Όταν βλέπουμε λοιπόν το γενικό συμφέρον και την παράβαση καθήκοντος και ποιος είναι ο ορισμός, οι διατάξεις υπάρχουν στην ε, νομοθεσία και η Ιρλανδική νομοθεσία και η Βρετανική το έχουν. Οπότε υπάρχει, μιλάμε για ποινικό αδίκημα, ε, κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια, ε, κακοδιαχείριση, κίνδυνο για την, ε, για την για τη δημόσια υγεία ή στραψοδικία. Μιλάμε δηλαδή για σοβαρές, σοβαρά εγκλήματα και βεβαίως πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο που να τα ρυθμίζει. Δεν, ε, ο προηγούμενος νόμος δεν τα κάλυπτε όλα αυτά και αυτό πρέπει να αλλάξει γιατί οποιαδήποτε διαφορά σε επίπεδο προσωπικού και ιεραρχίας έμπαινε σε αυτό το πλαίσιο. Οπότε χανόταν η αξιοπιστία ουσιαστικά αυτών των ε, κανόνων γιατί θεωρείται ότι για οποιοδήποτε ε, διαφορά υπήρχε μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου έμπαινε η ε, καταγγελία και οι κανόνες αυτές τις τιμές. Οπότε νομίζω ότι είναι αρκετά δύσκολο να περιμένουμε από ένα άτομο να καταλάβει απόλυτα το τι λέει ο νόμος. Βεβαίως ε, είναι δύσκολο να ξέρει κανείς και τι είναι το δημόσιο συμφέρον, αλλά εγώ αυτό που θέλω είναι να έχετε έναν κατάλογο που να δείχνει παραδείγματα ήδη αδικημάτων και να επιτρέπει στον νόμο να παρέμβει. Αν θέλουμε δηλαδή κάτι που να είναι κλειστό, τότε όσοι ασχολούνται με θέματα αφρολογικά ή με θέματα ηθικής δεν θα καλύπτονται. Πρέπει να πιστεύουμε αυτόν που κάνει την ε, καταγγελία. Και νομίζω ότι ω προ αυτό η προσέγγιση είναι καλή. Μιλήστε και για την ε, καλή πίστη. Και αυτό μα έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε τέτοιε ε, δικαστικές διαδικασίες, ε, γιατί μπορεί να μπορείτε να, μπορεί κάποιος να σας πει ναι, δεν, θα το, δεν το έκανε ε, αυτό με, την, ε, με καλή πίστη και προσπαθεί ο άνθρωπος να αποδείξει όντως ότι δεν είχε κάποιο απότερο συμφέρον για την καταγγελία που έκανε, αλλά όντως μόνο την καταγγελία θέλει να κάνει. Οπότε πρέπει να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που του δίνουμε προστασία και αν μπορεί η εταιρεία να αποδείξει ότι δεν ενέργησε καλόπιστα, τότε μπορεί να μειωθεί η αποζημίωση. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα όριο. Όταν μπαίνει κανείς μέσα σε μια τέτοια διαφορά και οι πληροφορίες δεν ε, τη χάνουν καλής μεταχείρισης και χάρη τη δουλειά σου επειδή κατήγγειλε αυτό που κατήγγειλε, μετά θα υπάρξουν προβλήματα. Προφανώ θα υπάρξουν και διαφωνίε, θα υπάρχουν γιατί όντω βρίσκεσαι σε μια προσπάθεια επίλυσης διαφοράς. Και εκεί αρχίζουν να, να, ε, να υπάρχει και ένταση στις ε, επαγγελματικέ σχέσεις. Αλλά συνήθως ε, ε, παραβλέπουμε αυτά που κάνουν άνθρωποι που, μας, που συμπαθούμε και συνήθως επικεντρωνόμαστε σε αυτά που κάνουν αυτοί που δεν συμπαθούμε. Οπότε είναι πολύ εύκολο να παραβλέψει κανεί αν καταγγέλλοντα. Και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει σαφής, ε, σαφές, εντό σαφής διατάξεις εντός της Νομίζω ότι απήντησα εγώ. Θέλετε να απαντήσετε και την ερώτηση για τους διαφορετικούς τρόπους για το αν γνωρίζει κανείς την καταγγελία αυτό, τι πρέπει να κάνει για να διευκολυνθεί κανείς στην, υποβολή μια καταγγελία. Εμεί δουλεύουμε πολύ σκληρά ώστε να γίνει καλύτερα αυτή η δουλειά από τι διάφορε οργανώσει, γιατί έτσι μπορεί να προωθηθεί το θέμα. Ένα από τα όσα κάναμε το 2013 ήταν μια έρευνα με την Επιτροπή περί καταγγελιών, με όλες τις πρακτικές, έτσι ώστε να προσπαθήσουν να βοηθηθούν, μάλλον οι οργανώσεις να προωθήσουν την υποβολή καταγγελιών. Όταν αυτό γίνεται στην, στο χώρο εργασίας, προφανώς πρέπει τα πράγματα να γίνουν σωστά. Είναι προ το συμφέρον όλων αλλά έχουμε και τα θέματα της ε, ε, νομικής, ε, της νομικής προστασίας, οπότε νομίζω το κοινό πρέπει να γνωρίζει τι ακριβώς γίνεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή και τους εισηγητές για τις ερωτήσεις σας. Πολλά στοιχεία και λίγος ο χρόνο, οπότε θα προσπαθήσω να απαντήσω. Αναφέρατε τις διαφορές που υπάρχουν στα κράτη-μέλη και όντως αυτό είναι το γενικό αίσθημα. Ε, πρέπει να δούμε βεβαίω και την ε, αρχή τη επικουρικότητα. Είναι νομική απέτηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό ακριβώ βοηθά στην ε, ενίσχυση τη νομική ασφάλεια που μπορείτε να προσφέρετε. Και αυτό με φέρνει σε κάτι που σχετίζεται άρρηκτα με αυτό που λέω. Ποια είναι η προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια θα, είναι, θα πρέπει να είναι. Αν έχουμε μια τομιακή προσέγγιση, θα ενισχύσουμε τον κατακαιρματισμό Οπότε ουσιαστικά είναι αντιπαραγωγικό σε σχέση με αυτό που θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουν τα κρατημένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο αντί να αυξήσουν την νομική βεβαιότητα και την προστασία για όλους. Και έρχομαι στο ερώτημα της νομικής βάσης. Εγώ ασχολούμαι τα τελευταία δύο χρόνια με το θέμα αυτό και υπάρχει μια ε, έκθεση η οποία ήδη έχει δημοσιευθεί πριν από ένα-δύο μήνες όπου συζητούμε ακριβώς το θέμα των εξουσιών που, θέσατε, που θέσατε και εσείς αλλά για την γενική συζήτηση τώρα αυτό που βλέπουμε σαφώς και στην ομολογία του δικαστηρίου είναι και συνθήκε βέβαια ότι οι υπονοούμενε ε, εξουσίε θα πρέπει να ε, βασίζονται σε κάτι που να υπάρχει στη συνθήκη. Πρέπει δηλαδή να υπάρχουν για να διευρύνουν το επίδειο ε, των αρμοδιοτήτων των εξουσιών που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν δούμε τι εξουσίε τη Ευρωπαϊκής Ένωση, έχουμε μια γενική λεπτομερή εικόνα μέσω των διαφορών άρθρων. Μιλούμε για θέματα ιστορική αγορά για θέματα προστασίας εργαζομένων. Ίσως ήδη να είναι διαφορετικό το σκεπτικό, αλλά ο στόχος είναι να προστατεύσουμε τους ε, καταγγέλλοντες εκεί που γίνεται η καταγγελία. Άρα η δημόσια, αν η δημοσίευση γίνεται στον ε, δημόσιο χώρο, ε, αυτό βασίζεται στο 114, 140 συγγνώμη, ή αν θέλουμε να ε, προστατεύσουμε τον εργαζόμενο ή τον καταγγέλλοντα ανεξάρτητα από το που κάνει την καταγγελία του. Και εκεί το 114 δεν το καλύπτει αυτό. Γιατί εκεί περιοριζόμαστε μόνο στον ιδιωτικό τομέα. Δεν μπορούμε να καλύψουμε και το δημόσιο τομέα και τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μια λεπτομερή συζήτηση σχετικώ, αλλά μπορώ ευχαρίστω να σα δώσω τι ε, νομικέ εφέσει που λάβαμε για το ποιε είναι οι αρμοδιότητε και ποια είναι τα, τα συν και τα πλήν κάθε νομική βάση. Για τι βέλτιστε πρακτικέ τώρα και τι χείριστε πρακτικέ, δεν θα ήθελα τώρα να δείξω με το δάχτυλο όλους αυτούς που δεν ε, δρούν σωστά, αλλά όπως είπατε στην πρώτη παρέμβαση, από το θέμα δεν είναι αν είναι η γραμμή ή αν είναι η νομοθεσία σωστή. Βλέπουμε κράτη που έχουν νομοθεσία, αλλά όπως είπε και η Κάθη, από την πρακτική οπτική, το θέμα είναι αν εφαρμόζονται αυτές, αυτοί οι νόμοι που υπάρχουν. Οπότε στην, ε, στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό που μπορούμε να αντλήσουμε το δίδαγμα δεν είναι μόνο σε αν νομικώ κάνουν καλή δουλειά τα κρατημέλη, είναι ποιε είναι οι πρακτικέ που μπορούν να ακολουθήσουν και που έχουν λειτουργήσει. Και αυτό μπορεί να γίνει και σε χώρε που δεν έχουν συγκεκριμένου κανόνε, όπω α πούμε η Δανία. Υπάρχουν διαδικασίε που μπορούν να πλησιώσουν τι καταγγελίε, παρόλο που δεν υπάρχει ε, αμυγή νομοθεσία για την προστασία των καταγγελόντων. Και για, τις, ε, για την αποζημίωση. Όντω, ε, τα κρατη που έχουν συγκεκριμένα, συγκεκριμένη νομοθεσία δεν έχουν κατά ανάγκη και κανόνες για την αποζημίωση. Και για τα κρατη που έχουν μόνο μερική προστασία, αν είναι, εξαρτάται αν είναι αστικού ή ποινικού δικαίου. Υπάρχουν διαφορετικές άγουσες ε, για, ε, για την ευθύνη και, τα, ε, ε και τις αξιώσεις κτλ. Οπότε αυτό μπορούμε να το δούμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επίπεδο παρόλο που συμμερίζομαι και τις, ε, τις ε, ανησυχίες της ε, προηγούμενης ομιλήτριας ότι θα πρέπει να δούμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο τι μπορούμε να κάνουμε σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις. Ε, αυτά τα έχω στείλει και γραπτός βεβαίως στις απαντήσεις μου στις ερωτήσεις σας, οπότε μπορείτε να τα δείτε. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ερωτήσεις οι οποίες είναι κάπως περίπλοκες σχετικά με τη νομική βάση και την θεωρία των αυτονόητων, αν θέλετε, αρμοδιοτήτων. Καταρχάς, σε σχέση με αυτές, για να υπάρξει μια τέτοια αρμοδιότητα πρέπει να υπάρχει και να προϋπάρχει μια βασική αρμοδιότητα. Και η εσωτερική αγορά έχει μια συνολική αντιμετώπιση του θέματος και όχι μια διατομεακή. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να ορίσουμε σωστά και τα όρια της ελευθερίας έκφρασης και στο συγκεκριμένο τομέα δεν υπάρχουν αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με γενικά το συγκεκριμένο τομέα. Και γι' αυτό ακριβώς ε, είχα θεωρήσει χρήσιμη την ρήτρα εφικτότητας εισαγωγικά στο εσωτερικό των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να αναφερθούμε επίσης και στις εργασίες των ε, κρατών μελών και, των, ε, και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εκεί δεν υπάρχει κάτι το οποίο να αναφέρεται άμεσα ε, στην ε, κατανομή των αρμοδιοτήτων. Τώρα για το βάρος της απόδειξης ε, θα πρέπει αυτό να ανήκει στις επιχειρήσεις, γιατί αλλιώς το σύνολο της έννοιας της προστασίας δεν θα έχει καμία βάση και τώρα στην περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί κακή πίστη καταγγέλλοντος, τότε μπορεί να υπάρξει ίσως αναστροφή του βάρους της απόδειξης. Τώρα, για τις υποχρεώσεις των κρατών μελών που θα μπορούσαν να επιβάλλουν μάλλον τα κράτη-μέλη και για την δυνατότητα ύπαρξης μιας οδηγίας δεσμευτικής δηλαδή. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την ιδέα της προστασίας του καταγγέλλοντος, όπως επίσης και με την βάση θα έλεγα κάποιων δικαιωμάτων τα οποία είναι αναφέρετα και έχουν ήδη συζητηθεί σε επίπεδο Συμβουλίου της Ευρώπης. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με την ιεράρχηση των διαδικασιών για να ξεκινήσει η καταγγελία. Εδώ πρέπει να αναφερθούμε στην ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και πάντα παραμένει το πρόβλημα το πώς θα αντιμετωπίσουμε ε, εξ αρχής την έννοια του καταγγέλλοντος και πώς εντάσσεται η έννοια αυτή στα πλαίσια της νομικής μας τάξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η κυρία Ροζιτάχη και θέλει να απαντήσει. Ναι, σας ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις συγκράτησα που έχουν να κάνουν με την εντολή της διαμεσολαβήτριας ε, και τους κανόνες ε, για ε, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά την εντολή, έχει θεσπιστεί στη συνθήκη και είναι αρκετά ευρεία. Η διαμεσολαβήτρια πάντα είναι διατεθειμένη να εξετάσει ιδέες διεύρυνσης της εντολής εφόσον έχει και το απαραίτητο δυναμικό. Ε, τούτη τη βδομάδα η διαμεσολαβήτρια έστειλε επιστολή στην ε, επόμενη την Εσθονική Προεδρία για μια προσπάθεια ε, από ό,τι φαίνεται για περιορισμό της εντολής της διαμεσολαβήτριας. Ε, έχουμε λοιπόν εδώ ακριβώς την αντίθετη περίπτωση. Είμαστε διατεθειμένοι να εξετάσουμε τις δυνατότητες διεύρυνσης της εντολής, αλλά δεν είμαι βέβαιη ότι αυτό είναι απαραίτητο αυτή τη στιγμή. Ε, Έχουμε τον κανόνα εξέτασης καταγγελιών όταν ο καταγγέλλον νιώθει ότι δεν τον έχουν πάρει στα σοβαρά ή αν έχει ε, αντιμετωπίσει αντίπεινα εντός του χώρου εργασίας του. Τέτοιου τύπου ε, καταγγελίες λαμβάνουμε στον τομέα αυτών, όχι πολλές όμως. Και αυτό, για να απαντήσω στον κύριο Σέση, μπορεί να συμβαίνει επειδή τα πράγματα λειτουργούν καλά εντό των θεσμικών οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αντιμετωπίζονται σωστά οι καταγγέλλοντε διαμαρτυρίε και δεν θεωρούν ότι είναι απαραίτητο να ε, μεταφέρουν τις περιπτώσεις τους, τις υποθέσεις τους στη διαμεσολαβήτρια ή μπορεί ε, να μην γνωρίζουν οι εργαζόμενοι τι πρέπει να κάνουν. Πέρα από τη δουλειά αυτή αναφερόμαστε ε, σαφώς στο άρθρο 22β ε, του, του καταστατικού για τους ε, υπαλλήλους. Όταν λοιπόν κάποιος έχει προσφύγει στον Όλαφ και έχουν περάσει 60 μέρες, μπορεί να έρθει σε εμά. Έχουμε λοιπόν συγκεκριμένο κανόνα για καταγγέλλοντες, αλλά δεν λαμβάνουμε πολλές αναφορές. Ίσως επειδή τα πράγματα λειτουργούν καλά ή επειδή επιλέγουν να στραφούν προς κάποιον εξωτερικό φορέα. Είμαστε ένας από τους ε, σαφείς ε, Είμαστε ένας από τους συγκεκριμένους φορείς που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή. Επίσης, κάτι που θα έπρεπε να είχα αναφέρει και που δεν ανέφερα είναι οι ανώνυμες καταγγελίες. Για παράδειγμα, η διαμεσολαβήτρια έλαβε ανώνυμη καταγγελία πριν δύο-τρία χρόνια σχετικά με πρώην επίτροπο. Ο καταγγέλων ισχυριζόταν ότι είχε παραβιάσει τον κώδικα δεοντολογίας των επιτρόπων. Η διαμεσολαβήτρια δεν γνώριζε για ποιον πρόκειται, οπότε ξεκίνησε δική της έρευνα πρωτοβουλίας. Αυτό λοιπόν είναι τρίτο είδος καταγγελίας που μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι εμπίπτει σε αυτόν τον γενικό ε, τομέα της καταγγελίας παρατύπιων. Προτού λοιπόν θέλετε να αλλάξετε την εντολή της διαμεσολαβήτριας, φροντίστε να γνωρίσετε τι ακριβώς ε, περιλαμβάνει. Η κυρία Γκράς, παρακαλώ. Ε, Όπως είπα νωρί, εμείς είμαστε υπέρ της δημιουργίας ενός πλαισίου. Το είδαμε σε ορισμένε γαλλικές επιχειρήσεις και θα ε, καταστούμε σύντομα συμβατή. Η ανησυχία που υπάρχει είναι να αφήσουμε στις επιχειρήσεις μια κάποια ευελιξία έτσι ώστε να δημιουργήσουν τα αποτελεσματικότερα των διαθέσιμων μέσων. Υπάρχουν όπως είπα διαφορετικού τύπου επιχειρήσεις, διαφορετικού μεγέθους ε, και εδώ υπάρχει ένα ρόλος τον οποίο καλείται να παίξει η επιχείρηση, να δημιουργήσει δηλαδή ένα σύστημα επικοινωνίας, ιδιαίτερα στις μεγάλες επιχειρήσεις και εργοστάσια, για την, ε, ε, για την κυκλοφορία αν θέλετε της πληροφορίας. Ε, υπάρχουν κάποια προβλήματα ερμηνείας μερικές φορές, υπάρχουν θέματα πρακτικά τα οποία τίθενται, ποιος αντιμετωπίζει σε μια πρώτη φάση ε, την καταγγελία, τι γίνεται με τον σεβασμό των ατομικών στοιχείων, εδώ υπάρχουν εντελώς διαφορετικές ρυθμίσεις ανά χώρα θα πρέπει επίσης να δημιουργήσουμε ή μάλλον να πάρουμε κάποια μέτρα τα οποία να εγγυώνται ακριβώς το απόρριτο αυτής της επικοινωνίας. Αυτό το οποίο είχαμε στο παρελθόν ήταν να υπάρχουν άτυπες μορφές ενημέρωσης, ε, κάποιες επιχειρήσεις. Μερικές φορές ε, είναι αποτελεσματική αυτή η άτυπη επικοινωνία, αλλά δεν εγγυάται πάντα τις απαιτήσει ε, του νόμου ΣΑΠΑΝ 2 για την προστασία του απορρίτου και των ατομικών του στοιχείων και γεγονότων. Δεν εγγυώνται επίσης και μια χρονική προθεσμία αντιμετώπισης της καταγγελίας. Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε να είμαστε κατά της άτυπης διαδικασίας καταγγελίας, αλλά θα πρέπει να δώσουμε την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν ένα μέσο εσωτερικό αντιμετώπισης των καταγγελιών, να έχουν μια αποτελεσματική μορφή επικοινωνίας έτσι ώστε να ενημερώνονται οι μισθωτοί, οι εργαζόμενοι για την ύπαρξη των διαθεσίμων μέσων, για τον χρόνο και τα στάδια αντιμετώπισης της καταγγελίας, προθεσμία εννοώ, και να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να δημιουργήσουν, αν θέλετε, τα εσωτερικά συστήματα τα οποία απαιτούνται από πλευράς τους. Μια τελευταία παρατήρηση. Δεν είμαστε ε, υπέρ το να υπάρχει θα έλεγα μία άμεση καταγγελία σε σχέση με τους ανώτερους ιεραρχικά. Αυτό μπορεί να είναι εντελώς προσωπικό Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει επίσης ε, ένας, ε, ένα, ένα κομμάτι του προσωπικού που να ασχολείται με τα θέματα αυτά, διευκολύνει την επικοινωνία. Έχω άλλους 7 ομιλητές, 7 μέλη και γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω. Ας ακούσουμε λοιπόν τις 7 αυτές ερωτήσεις και μετά να δώσετε απαντήσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να σεβαστούμε τον χρόνο που έχουμε στην διάθεσή μας. Ο πρώτος ομιλητής είναι ο Πασκουάλ Δεγράντες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τις ομιλήτριες. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλή ιδέα η συνάντηση αυτή, τον κοινό, την κοινή συνάντηση των δύο επιτροπών γιατί ασχολούμεθα πραγματικά με ένα θέμα το οποίο έχει τεράστιο πολιτικό βάρος και δεν θα πρέπει να υπάρχουν μόνο κάποιες αυθόρμητες θα έλεγα πρωτοβουλίες αλλά θα πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα εγγυήσεων στον τομέα αυτό. Άκουσα πολλά και ενδιαφέροντα από τις ομιλήτριες, άκουσα και κάτι συγκεκριμένο το οποίο μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο. Η αναστροφή του βάρους της απόδειξης σαν κανόνα είναι κάτι το οποίο είναι μάλλον λανθασμένο. Και α, ακούγοντας ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να ανοίγει και στην ιδιωτική σφαίρα και ότι θα πρέπει το βάρος της απόδειξης να πίπτει πάντα στον εργοδότη είναι κάτι το οποίο νομίζω δεν θα μας βρει σύμφωνος. Αυτό λοιπόν το θέμα της αντιστροφής του άκθους της απόδειξης ε, μπορεί να υπάρξει μόνο σε σχέση με συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου ο στόχος δικαιολογεί αν θέλετε τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται. Δύο επιπλέον σημεία σύντομα. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση της κοινή γνώμης και εμείς ε, η κοινοβουλευτική μας επιτροπή ε, ασχολείται με θέματα τα οποία προκαλούν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον της κοινή γνώμης. Ασχολούμεθα με συμπεριφορές ε, δεοντολογικές, νομικές που επηρεάζουν πάρα πολύ την πολιτική κατάσταση. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει βέβαια μια ατελείωτη νομιμοποίηση θα έλεγα να περάσουμε από το συγκεκριμένο θέμα και να προαποφασίζουμε εμείς το σε ποιον θα εμπίπτει το βάρος της απόδειξης, σε ποιο φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι το ισχυρισμό αυτός δεν είναι κάτι το οποίο με πείθει. Τώρα, ο ορισμός του καταγγέλλοντος. Υπάρχουν διαφορετικές νομικές ρυθμίσεις και αντιλήψεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα και με αυστηρότητα. θα πρέπει να μπορέσουμε να περιγράψουμε το συγκεκριμένο αυτό πρόσωπο. Τελειώνω λέει ο κ. Δεγκράντης. Δεν θα πρέπει να κάνουμε ένα σύστημα το οποίο να είναι απόλυτα δεσμευτικό, αλλά ούτε και ένα σύστημα απόλυτα φιλελεύθερο. Είναι αλήθεια ότι στο εσωτερικό των επιχειρήσεων οι συνδικαλιστικές αντιπροσωπευτικές οργανώσεις βρίσκονται σε παρακμή θα έλεγα, σε πτώση και θα πρέπει να υπάρχουν ε, δυνατότητες για τους εργαζομένους να καταγγέλουν απαράδεκτες πρακτικές. Είμαι υπέρ του να υπάρχουν, αλλά όχι θα έλεγα με αντιλήψεις οι οποίες προϋποθέτουν και επιβάλλουν συγκεκριμένες ιδέες δικαίου. και Σας ευχαριστώ για όλες τις ε, παρουσιάσεις αυτές. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να παρευρεθώ ε, ήδη από την αρχή λόγω σημαντικής ψυχοφορίας ε, στην Επιτροπή Πολιτισμού. Έχω όμως τις εξής παρατηρήσεις. Για την ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών είναι σαφές ότι οι κατακέλλοντες παίζουν σημαντικό ρόλο καταγγέλλοντας ε, παρατυπίες ε, και παράνομες δραστηριότητες. Είναι λοιπόν σημαντικό να διαφυλάξουμε το δημόσιο συμφέρον, να διασφαλίσουμε την διαφάνεια, να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο ε, έγκλημα και την φοροδιαφυγή. Αποτελούν λοιπόν σημαντικό πυλώνα στον αγώνα κατά της διαφθοράς και για την λογοδοσία των οργανισμών και επιχειρήσεων έχει έρθει η ώρα να προστατεύσουμε νομικά τους καταγγέλλοντες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ στο παρελθόν ε, το Κοινοβούλιο έχει πιέσει αρκετά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει υποβάλει ακόμα πρόταση. Όταν διώκεται δικαστικά ο καταγγέλλον, ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις ε, μπορούν να ε, φοροδιαφεύγουν και να φοροαποφεύγουν χωρίς κυρώσεις, ε, αυτό σημαίνει ότι κάτι πάει στραβά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρώτη μου ερώτηση είναι λοιπόν, βλέπετε συγκεκριμένα σημεία αναφοράς για την προστασία καταγγελόντων στις συνθήκες. Η κυρία Περό ήδη το εξήγησε αυτό. Υπάρχουν όμως και άλλα σημεία ε, αναφοράς. Δεύτερη ερώτησή μου. Ενώ θέλουμε να προστατεύσουμε τους καταγγέλλοντες, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε κλίμα φόβου και ε, απόσταση ανάμεσα στους εργοδότες και τους εργαζομένους ε, στις επιχειρήσεις. Χρειαζόμαστε σαφή διάκριση ανάμεσα στην καταγγελία ε, και στην κατηγορία συκοφαντία. Στο παρελθόν επίσης υπήρχαν διάφορες περιπτώσεις όπου εργαζόμενοι ελβετικών τραπεζών πούλησαν πληροφορίες σε αρχές ε, στην Γερμανία. Στην... Απ' τη μία ε, το πρόσωπο αυτό ε, έλαβε αμοιβή γι' αυτό, άρα εργάστηκε για προσωπικό του συμφέρον. Από την άλλη όμως ήταν για το δημόσιο συμφέρον. Ένα τέτοιο πρόσωπο θεωρείται καταγγέλων, πρέπει να προστατεύεται νομικά. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρουανελέν, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τις ε, εμπειρογνώμονες για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις τους. Φυσικά πρέπει να προστατεύσουμε του καταγγέλλοντε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναρωτιέμαι όμω η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα κατάλληλα μέσα για να βελτιώσουμε την προστασία καταγγελόντων και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, Για παράδειγμα, σε περιπτώσει συγκρίσιμε με την περίπτωση των εγγράφων του Παναμά τι γίνεται αν αποκαλυφθεί η, η ιδιότητα του καταγγέλλοντος και διωχθεί δικαστικά το πρόσωπο αυτό στον Παναμά. Έχουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσουμε και τέτοιες περιπτώσεις ή μπορούμε να αναπτύξουμε τα απαραίτητα μέσα. Τις τελευταίες δεκαετίες ε, είδαμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για, τις, ε, για τους κανόνες των επιχειρήσεων και τα Ηνωμένα Έθνη όπως και όσα έχουν εκπονήσει κώδικα δεντολογίας για πολυεθνικές επιχειρήσεις. Πιστεύετε ότι τέτοιες κατευθυντήριες γραμμέ αποτελούν δυνατότητα για βελτίωση τη προστασία των καταγγελόντων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Ε, en primer lugar, el agradecimiento a todas ustedes. Βρισκόμαστε εδώ γιατί σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο και με την τεχνολογική επανάσταση, πάρα πολλά φαινόμενα διαφθοράς, παρανομίες κτλ. είναι διεθνικού χαρακτήρα. Και εμείς σαν βουλευτές προσπαθούμε να τοποθετηθούμε απέναντι σε αυτό για να προστατεύσουμε τους καταγγέλλοντες καταστάσεις δημοσίου συμφέροντος. Η κυρία Χίκη, η τελευταία μιλήτρια, είπε ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε το πότε και πόσο γίνεται η καταγγελία. Τίθεται επίσης και το θέμα της νομικής βάσης, το 114 και το 352. Το θέμα είναι να αναγνωρίσουμε ακριβώς ότι πρέπει να υπάρχει ελευθερία έκφρασης. Θα πρέπει να αναγνωριστούν φυσικά οι δυνατότητες των δικτύων των διαμεσολαβητών κάτι το οποίο δεν είναι πάντα εφικτό. Πώς λοιπόν μπορούμε να έχουμε μία νομική βάση η οποία θα έλεγα μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνολικά. Να επιβάλλει αν θέλετε μία κουλτούρα α, και στον ιδιωτικό και στον, και στον δημόσιο τομέα για την προάσπιση της δημοκρατίας. Θα πρέπει επίσης να προσπαθήσουμε να αναγνωρίσουμε και τα όρια της εμπιστευτικότητας στον τομέα αυτό και πώς μπορεί να στραφεί επίσης και στις υπηρεσίες του διαμεσολαβητή ένας καταγγέλων. Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετές απορίες πάνω στις οποίες και οι δύο μας επιτροπές μπορεί να χρησιμοποιήσουν για να εργαστούν ορθότερα. Από την ΚΟΕ, ο κύριος Κρέσπο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις σας. Νομίζω ότι το θέμα αυτό έχει κεντρικό χαρακτήρα. Εμείς αν δεν υπήρχαν καταγγέλλοντες δεν θα γνωρίζαμε τα έγγραφα του Παναμά και δεν θα υπήρχε η Επιτροπή μας. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τον ρόλο των καταγγελών, των ανδρών και γυναικών Αλλιώς δεν θα γνωρίζαμε διάφορα σκάνδαλα στην Ισπανία όπως των οικονομικών του Λαϊκού Κόμματος, δεν θα γνωρίζαμε τον Ασάνζ και άλλες περιπτώσεις και ε, πληροφορίες γύρω από τον πόλεμο του Ιράκ, γύρω από τα Λουξ λίξ και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει μια νομοθετική ρύθμιση η οποία να προστατεύει τους καταγγέλλοντες ως προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και γι' αυτό θα ήθελα να σας θέσω κάποιες ερωτήσεις και κάποια στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να διευκολύνουν την συζήτηση την οποία θα έχουμε ε, για τα ε, έγγραφα του Παναμά. Καταρχάς, σε τι εμπειρίες ε, ε, πραγματικά ενδιαφέρουσες μπορούμε να στραφούμε για την προστασία ε, των, των καταγγελόντων που θα μπορούσαν να εξαχθούν, θα έλεγα, σαν βέλτιστες πρακτικές σε άλλες χώρες. Που θα μπορούσαν λοιπόν να χρησιμοποιηθούν και αλλού και προς την κατεύθυνση αυτή πώς είναι δυνατόν να εφαρμοστούν αυτές οι, οι αντίστοιχες εμπειρίες, όχι μόνο να γνωρίζουμε αλλά και να αναπαράγουμε. Πώς επίσης μπορούμε να αναπαράγουμε ε, βέλτιστες πρακτικές και στο εσωτερικό των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ε, πιθανώς θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως ε, ε, καταγγέλλοντες. Τι μέτρα χρειάζονται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρω ότι επικοινωνούμε με τον Ασάνζ. Τι ιδέες μπορούμε να πάρουμε έτσι ώστε να φτιάξουμε κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά ακόμα και πέραν αυτής και για την οδηγία τώρα για τα επιχειρηματικό απόρριτο, την οποία εγκρίναμε τον Απρίλιο του 2016, η οποία υφίσταται κριτική και η οποία θα έλεγα χειροτερεύει και δυσκολεύει τον ρόλο των καταγγελόντων και εμείς ε, πραγματικά είχαμε πει ε, να περιμένει η οδηγία αυτή, να ε, κλείσει η ιστορία του ελέγχου των εγγράφων του Παναμάτ και μετά να περάσουμε στην επόμενη οδηγία, αλλά κάτι το οποίο δεν έγινε. Έχω και άλλες ερωτήσεις, δεν έχω όμως χρόνο. Περιμένω με ενδιαφέρον τις απαντήσεις σας. Σας ευχαριστώ. Σκοτ Κέιτο. Θα ήθελα να επανέλθω σε αυτά τα οποία είπε ο πρόεδρος Χαίρομαι που βλέπω ότι είστε όλες εδώ γυναίκες. Θυμάμαι αυτό που είχε πει ότι ο Μπένετ, ότι οι γυναίκες ακολουθούν τους άνδρες μαζί με ένα κουβά για να μαζεύουν τα λάθη τους. Λοιπόν, και το πρώτο, η πρώτη παρατήρηση αφορά το βάρος της απόδειξης. Ε, εμείς προετοιμάζουμε μια γνωμοδότηση στην ΕΚΟΝ για την αντιστροφή του βάρους της απόδειξης και προσπαθούμε να βρούμε κάποιες λύσεις στα προβλήματα που υπάρχουν. Δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωμένοι οι καταγγέλλοντες να αποδείξουν ότι το κάνουν αυτό που κάνουν καλή την πίστη, ακόμα και αν υπάρχουν κάποιες ανακρίβειες και θα πρέπει ο εργοδότης, όπως είπατε, να αναλαμβάνει το βάρος της απόδειξης. Πώς είναι δυνατόν να βρούμε μια διατύπωση η οποία να αντιπροσωπεύει την πραγματική ε, θέση του βάρους ε, της απόδειξης και πώς ε, η θεωρία γύρω από το βάρος της απόδειξης δεν είναι αρρωγός των προσπαθειών που κάνουν οι καλαγγέλλοντες στην παρούσα φάση ενώ υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν καταφέρνει κάποιος να αποδείξει ότι ε, το κάνει για το κοινό συμφέρον, ενώ είναι σαφές ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει. Εμείς στην ε, πράσινη πρόταση που είχαμε κάνει για την προστασία των καταγγελόντων, είχαμε μιλήσει για τη χρήση του άρθρου του 153 και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Έχει σημασία εδώ αυτό το οποίο είπατε για την έλλειψη ισορροπίας ε, ανάμεσα στους εργαζομένους και τους εργοδότες. Ένας λόγος είναι η ε, απίσχναση θα έλεγα της παρουσίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων και πώς μπορούμε τελικά να χρησιμοποιήσουμε τη συνθήκη για να βοηθήσουμε τους καταγγέλλοντες. Αν έχω κάποιες πληροφορίες από ένα πρόσωπο για μια μεγάλη επιχείρηση, πώς είναι δυνατόν να έχω ένα πλαίσιο νομικό που θα του επιτρέψει να κάνει ένα ακόμα βήμα και να δημοσιοποιήσει αυτά τα οποία ισχυρίζεται. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ εγώ που είναι μόνο γυναίκες ευρωγνώμονες σήμερα εδώ. Ένα μήνυμα ήταν πολύ σημαντικό. Να πούμε ότι χρειαζόμαστε τους κατακέλλοντες. Κυρίως για την ε, διαφορά, για την φοροδιαφυγή. Όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, κακοδιαχειρήσεις ε, στα κρατημέλη, είναι σημαντικοί οι καταγγέλλοντες. Και μάλιστα μία εμπειρογνώμων είπε ότι είναι δημοκρατικοί παίκτες. Η Κομισιόν τον Μάιο μας ζήτησε να τις πούμε ποιες είναι οι δυνατότητες προστασίας στο, των καταγγελόντων. Κοίταξα εγώ τα κείμενα ε, για την αποφυγή ας πούμε της ποινικής δίωξης είναι πολύ ενδιαφέρον όμως να λέμε ότι θα πρέπει να βρεθεί μια γενική υπερεθνική λύση. Αυτή η παράγραφος 114. Μία μα ε, είπε ότι αυτό αρκεί μόνο όταν έχουμε μία διεύρυνση του τρέχοντο πεδίου εφαρμογή. Νομίζω όμω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουμε κανόνες που να μπορούν να γίνουν αποδεκτοί και από τα κράτη-μέλη. Οι υπόλοιποι πώ το βλέπουν αυτό. Και επίση, άλλο ένα σχόλιο. Ένα καταγγέλων μπορεί να κάνει ας πούμε μια θηρίδα δική του ώστε να μην δημοσιεύεται η διεύθυνσή του ώστε να μην υπάρξει δυνατότητα ποινική του δίωξη. Είναι δυνατό αυτό ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλειά του. Θα με ενδιαφέρει αυτό. Ευχαριστώ. Now, ε, να ακούσουμε τις απαντήσεις. Έχουμε τον κατάλογο των ομιλητών. Θα ακούσουμε τις απαντήσεις και μετά θα κάνουμε ένα catch the eye. Uh, we are uh, Κυρίες μου, δεν έχουμε πολύ χρόνο, οπότε έχετε το υπόψη σας αυτό όταν θα απαντήσετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα ερωτήματά σας. Εγώ είμαι η δικηγόρο νομικό τη υπόθεση, οπότε θα αφοσιωθώ στα νομικά και μπορώ βεβαίω να κάνω και κάποια σχόλια για τα υπόλοιπα ερωτήματά σα, αν θέλετε. Ένα από τα σημεία που συζητάτε συνεχώ και αναφέρεται από όλου όσου παρανέβησαν είναι το θέμα τη νομική βάση. Ποια είναι η νομική βάση που θα χρειαστούμε και ποιοι είναι οι περιορισμοί. Για να το πω απλά, αν χρησιμοποιήσουμε το 114 τη συνθήκη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ρυθμίζει την ιστορική αγορά, σημαίνει ότι περιορίζουμε την προστασία των καταγγελόντων στον ιδιωτικό τομέα. Το καλό τη χρήση αυτού του άρθρου, όπω είπα πριν, είναι ότι μπορεί να παράσχει ένα μέτρο που θα ζητά από τα κράτη-μέλη να εναρμονίσουν την προστασία που παράσχουν. Οπότε ζητά περισσότερα από τα κρατημένες ό,τι αφορά τι δράσει του για την προστασία των καταγγελόντων. Αλλά το ερώτημα πάλι που τίθεται είναι αν θεωρούμε ότι είναι ικανοποιητική αυτή η προσέγγιση. Γιατί θα ενισχύσει τον καταγγελματισμό αντί να τον ε, ε, διορθώσει, γιατί αφήνει σημαντικά, σημαντικές πτυχές εκτός προστασίας των καταγγελόντων. Το άρθρο 114 θα μπορούσε δυνητικά να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την προστασία τη υγεία ή του περιβάλλοντο, που δεν είναι και ασύνηθε, ε, σε ό,τι αφορά τα όσα προκύπτουν από διάφορες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και πάλι είναι θέμα πεδίου εφαρμογής. Ε, το 153 ε, ίσως να είμαι λίγο ε, ε, προκατηλημένη γιατί ε, ήμουνα μία από τις συντάκτριες της σχετικής νομοδότησης. Το άρθρο αυτό καλύπτει ακριβώς τον εργαζόμενο, το άτομο, ανεξάρτητα από τη θέση που έχει, από τον τομέα που δουλεύει, από το που βρίσκεται. Ανοίγει λοιπόν έτσι ο δρόμος των, ε, της προστασίας για όλα τα είδη των καταγγελόντων. Οπότε θέλω να υπενθυμίσω σε όλους το παράδοξο που υπάρχει και που αντιμετωπίζουν οι καταγγέλλοντες στην Ευρώπη σήμερα. Συχνά θέλουν να συχνά κάποιοι ε, φυλακίζονται στην χώρα τους, συμβάνονται στη χώρα τους, ενώ την ίδια χρονιά το κοινοβούλιο, ας πούμε, τους ε, διακηρύσει πολίτε της χρονιάς επειδή διαφυλάσσουν τη δημοκρατία. Οπότε πρέπει να δούμε αν θέλουμε να συνεχίσουμε και στο μέλλον να αφήνουμε ανοιχτό αυτό το παράδοξο ή αν πρέπει να βρούμε κάποια νομική ε, βάση που θα μπορέσει να καλύψει το πρόβλημα. Για το βάρος της απόδειξης, η νομική πρακτική δείχνει γιατί υπάρχουν χώρε όπω είπα που έχουν προστασία, κανόνε για την προστασία εδώ και δεκαετίε των καταγγελόντων. Τη στιγμή λοιπόν που το βάρο εναπόκειται στον ε, καταγγέλλοντα, ε, ουσιαστικά αντί, αντιφάσκει με την, με την όλη ιδέα της καταγγελίας. Οπότε συμφωνώ με αυτά που είπαν οι προηγούμενοι ότι μπορούν να γίνουν κάποιες διακρίσεις εδώ μεταξύ της προστασίας. Η προστασία θα πρέπει να υπάρχει καθ' αυτή, ενώ η αποζημίωση μπορεί να υπόκειται σε κάποιες προϋποθέσεις ε, καλής πίστης ας πούμε κτλ. ή ε, εύλογης ε, ε, αξιοπιστίας των λεγόμενων. Νομίζω ότι Α, κάτι άλλο που ετέθη είναι το θέμα της εφαρμοσιμότητας του νόμου εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι γίνεται δηλαδή αν κάποιος κατηγορείται σε άλλο κράτος. Γενικώ θα υπάρξει μια παρακολούθηση σε ό,τι αφορά την, ίσως την ε, ε, εθνικότητα του ατόμου και μπορεί ίσως να βρεθούν κάποια ένδικα μέσα στη χώρα τη καταγωγής του και όχι στη χώρα της δημοσίευση της καταγγελίας. Γιατί όπως υπόθηκε πολλέ από τις καταγγελίες είναι ε, υπερεθνικές. Οπότε πάντα θα υπάρχουν περισσότερες χώρες που τις αφορά. Και τέλος, ετέθη ένα ερώτημα για το κατά πόσο μπορούμε να έχουμε μια διεύθυνση ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν ε, οι ε, καταγγέλλοντε για να προστατεύσουν την ιδιωτικότητά του. Υπάρχουν τέτοιου είδου πρωτοβουλίε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω το Σεπτέμβριο του 2016 έγινε κάτι τέτοιο. Υπάρχουν πλατφόρμες ε, καταγγελόντων που λαμβάνουν όλο και περισσότερο προσοχή από τα ΜΜΕ. Αλλά βεβαίω. Πρέπει να υπάρχει η ε, ανωνυμία και πρέπει να μπορούν να ε, καταγγέλουν και να υποβάλουν τα έγγραφα που, τα σχετικά χωρίς να ε, διακυβεύεται η ανωνυμία τους. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη αν μακρηγόρησα. Πολλά σημεία έχουμε να καλύψουμε, αλλά πολλές καλές ερωτήσεις για την ανωνυμία. Αυτό θα το διαλέξει κάποιος αν, θεωρήσουν, ότι δεν είναι ασφαλής. Αν θέλουμε τώρα να έχουμε προστασία, σε κάποιον που βρίσκεται σε μια εταιρεία που δεν, ε, έχει, που δεν σκοπεύει να κάνει κάτι, θα πρέπει να δούμε πώ ε, μπορούμε αυτό να το αντιμετωπίσουμε. Και βεβαίω να δούμε και τι γίνεται με τι ερωτήσεις, με τις εταιρείε που θέλουν κάτι να κάνουν, Και εξαρτάται από το τι, ποια είναι η εταιρεία για την οποία δουλεύουν, τι είναι αυτό που θέλουν να αποκαλύψουν. Οπότε δεν είναι πάντα προφανέ να να έχουμε προστασία για ανώνυμη καταγγελία, γιατί αυτό σημαίνει ότι έχετε δώσει κάποιες πληροφορίες και έχετε, έχετε υποφέρει από κάτι, έχετε πληγεί με κάποιο τρόπο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κοιτάξουμε τρόπους που μπορεί κανείς ανώνυμα να κάνει μια καταγγελία. Γίνεται μεγάλη έρευνα από την ACCA στο Ηνωμένο Βασίλειο που μιλά ακριβώ για αυτά τα αυτέ τι διαφορετικέ προσέγγισει και τα είδη καταγγελιών που μπορεί να κάνει κάποιο έτσι ώστε να υπάρξει εμπιστοσύνη. Όλες αυτές οι άγουσες βεβαίως ε, άλλο το χρησιμοποιούνται πολύ και άλλο τα λίγο. Οπότε είναι δύσκολο να βάλουμε ένα νομικό πλαίσιο, αλλά είναι βεβαίως σημαντικό ότι για το βάρος της απόδειξης ο εργοδότης είναι αυτός που, κάνει την, που παίρνει την απόφαση να πωλήσει τον εργαζόμενο, να υπονομεύσει τη θέση του. Οπότε έχει νόημα να πρέπει αυτός να αποδείξει ότι υπήρχαν άλλοι λόγοι για τη δράση του καταγγέλλοντος. Οπότε δεν μπορώ να δω πώ πώς, μπορεί να έχει κάποιος άλλος το βάρος απόδειξη και όχι ο εργοδότης. Ο, ο καταγγέλλον λέει ότι έδωσε τις πληροφορίε και ε, υπέστην ε, κάποια βλάβη. Ε, οπότε ο εργοδότης πρέπει μετά να αποδείξει τι ήταν αυτό. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί τρόποι με τον οποίο μπορεί να προχωρήσει αυτό, εφόσον όμως έχει αναλυφθεί ο, το βάρος απόδειξη από τον εργοδότη. Το σημείο εκείνη όμως πρέπει να είναι ότι το βάρος απόδειξης εμπίπτει στον εργοδότη. Ε, για τα Panama Leaks, ναι πρέπει να έχουμε και έναν ένα μηχανισμό ε, προστασίας του δημοσίου συμφέροντος σε κάθε χώρα. Θα πρέπει να μπορούμε να αμφισβητήσουμε το τι γίνεται με τις καταγγελίες των ε, ε, ατόμων αυτό. Μιλάμε ας πούμε για ε, παραβίαση των, των απορρίτων. Πρέπει να υπάρχει κάποιο είδος προστασία. Και εκεί μιλάμε για την προστασία του καταγγέλλοντο, α πούμε, για την περίπτωση του Παναμά. Θα έπρεπε να μπορεί να παρουσιάσει ότι ήταν τόσο σημαντικέ για το δημόσιο συμφέρον αυτέ οι πληροφορίε, ώστε να μπορεί να υπερμενθεί τη υπόθεσή του, του εαυτού του ουσιαστικά, σε τέτοιε δικαστικέ διαδικασίε. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί που μπορούμε να σκεφτούμε σε ό,τι αφορά την πολιτική και όχι τόσο την νομοθεσία, για να μπορέσει όλο αυτό λειτουργικά να, ναι, πρακτικά να λειτουργήσει. Υπάρχει, υπάρχει μια δέσμη ε, αρχών για την ελευθερία του λόγου και υπάρχουν και σημεία επαφής ε, σε όλο το σύστημα υγείας για, την, ε, για τους καταγγέλλοντες. Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις που πρέπει να ακολουθήσουμε, αλλά βεβαίως πρέπει να υπάρχει κάποιος με γενική ευθύνη επιχειρησιακά και με γενική ευθύνη ε, πολιτικά σε εισαγωγικά. Ε, νομίζω ότι θα κλείσω εδώ γιατί μάλλον ε, χρησιμοποίησα περισσότερο χρόνο από ό,τι έπρεπε. Για το σύνολο των θεμάτων που άπτονται της νομικής βάσεως. Το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε είναι το τι θέλει να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να δημιουργήσει μια οδηγία δεσμευτική δηλαδή για τα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα στον τομέα της μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία, νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη λύση σε επίπεδο νομικής βάσεως πέραν αυτών που υπόθηκαν, εκτός και αν ξεκινήσουμε να βλέπουμε το θέμα τομεακά. Αν η ουσία είναι να προστατεύσουμε τους καταγγέλλοντες γιατί σαν παράδειγμα είναι απαραίτητο για την καταπολέμηση της διαφθοράς τότε μπορούμε να κάνουμε τομεακές ρυθμίσεις με κίνδυνο βέβαια να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τη διαφορετικότητα των αντιμετωπίσεων του θέματος. Το θέμα της κατανομής των αρμοδιοτήτων είναι το μοναδικό θέμα που μένει σε εκκρεμότητα σε νομικό επίπεδο και είναι κάτι το οποίο θα θέσει κινδύνο αν θέλετε μία νομοθετική ρύθμιση ευρύτερου πεδίου και που θα μπορούσε να αμφισβητηθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για νομικά κενά και λάθη. Κάτι το οποίο θα καθυστερήσει ακόμα περισσότερο την έβρεση μιας λύσης. Αν θέλουμε να προστατεύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα βλέπει τον καταγγέλλοντα ως ε, ε, πρωταγωνιστή της δημοκρατικής διαδικασίας, εγώ καταλαβαίνω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βλέπει το θέμα αυτό αρκετά περίπλοκο, γιατί το θέμα του βάρους της απόδειξης δεν είναι τόσο σημαντικό, αλλά θα πρέπει, θα έλεγα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημοσιοποιήσει μια σειρά προτάσεων, κατευθυντηρίων γραμμών, που θα ορίζουν το βάρος και τη σημασία του καταγγέλλοντα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση το θέμα της κατανομής των αρμοδιοτήτων σε επίπεδο νομικής βάσεως δεν τίθεται με τον ίδιο τρόπο. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο θα πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε λίγο είναι το τι θέλουμε να κάνουν τα κράτη-μέλη. Θέλουμε όλα τα κράτη-μέλη να περάσουν σε ένα επίπεδο προστασίας ή θέλουμε τα κράτη-μέλη σιγά σιγά να μπορέσουν να περάσουν σε μια ήπια εναρμόνιση των νομοθετικών τους ρυθμίσεων από τον τομεακό στον οριζόντιο, από μια πιο σημαντική προστασία από αυτή που προβλέπεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Εδώ θα πρέπει να δημιουργήσουμε κάποιες διαδικασίες σχετικές με την δημοσιοποίηση των εθνικών νομοθετικών ρυθμίσεων και θα πρέπει να δούμε εδώ τον ρόλο του διαμεσολαβητή έτσι ώστε να μπορέσουμε να ορίσουμε τις διαφορές, να ορίσουμε τις αποκλίσεις και τα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν μια περισσότερο κοινή αντιμετώπιση. Αυτή η αντιμετώπιση έχει θετικά στοιχεία και το συζητάμε σε ορισμένα θέματα. Είναι λιγότερο δεσμευτική για τα κράτη-μέλη το ερώτημα το οποίο τίθεται όμως είναι το τι έχει προτεραιότητα. Είναι ο εξαναγκασμός των κρατών μελών ή η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν ζώνης προστασίας, μία ζώνης προστασίας του καταγγέλλοντα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Χική. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά την ανωνυμία και την προστασία των καταγγελόντων καθώς και το βάρος απόδειξης στην ερώτησή σας. Ναι, πράγματι, όσον αφορά την ανωνυμία, λέμε ε, στον κόσμο, εάν θέλετε να απευθυνθείτε ανώνυμα στον, ε, στη διαμεσολαβήτρια, μπορείτε να το κάνετε, τότε όμως δεν προστατεύεστε. Όσον αφορά το βάρος της απόδειξης, θέλουμε να αποφύγουμε κάποια σενάρια. Δεν νομίζω ότι προσπαθεί κανείς να υπερασπιστεί το ε, σενάριο όπου οποιοδήποτε μπορεί να πει οτιδήποτε στον τύπο, να πρέπει η επιχείρηση να ε, ε, υπερασπιστεί τη θέση της και να έχει προστασία ο καταγγέλων. Εάν όμως πάρετε το παράδειγμα ενός ατόμου που δεν γνωρίζει εάν ε, αυτό που θέλει να καταγγείλει είναι παρκώς σοβαρή η παρατυπία, τότε φυσικά θα πρέπει να προστατεύεται. Δεν επιτρέπεται να μην προστατεύεται επειδή διαπιστώθηκε ότι αυτό που κατέγγειλε ε, δεν ήταν αρκετά σοβαρό και δεν εμπίπτει στο άρθρο 22 του ε, καταστατικού για τους ε, υπαλλήλους. Φυσικά σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να προστατεύεται το άτομο. Αλλά η προστασία δεν είναι χωρίς περιορισμούς και θα πρέπει να υπάρχει κάποιο άρθρο σχετικά με κατάχρηση της διαδικασίας ώστε να μην ε, πετάει κανείς κατηγορίες για διαφόρους για λάθος λόγους και να έχει ο εργοδότης το βάρος της απόδειξης. Όσον αφορά την ερώτησή σας σχετικά με το τι ρόλο μπορεί να παίξει ε, η διαμεσολαβήτρια, ο Όλαφ είναι το γραφείο καταγγελιών, διότι αυτό αναφέρεται μαζί με το δικό σας θεσμικό ε, όργανο. Πρώτα δηλαδή ε, καταγγέλει κανείς εσωτερικά και αν δεν έχει αυτό αποτέλεσμα απευθύνεται στον Όλαφ. Και ω δεύτερο επίπεδο πια έχει κανεί ε, τη διαμεσολαβήτρια, τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου και το ελεγκτικό συνέδριο. Μία από τις ε, καινοτομίες ε, στο νέο καταστατικό ήταν ότι αναφέρονται κανόνες, όχι πολιτικές, που μπορούν να εφαρμοστούν. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Γκράς. Να επανέλθω στην διάκριση ανάμεσα στην ανωνυμία και την εμπιστευτικότητα. Έτσι κι αλλιώ να αντιμετωπιστεί μια ανώνυμη καταγγελία σε μια επιχείρηση είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν μπορούμε πώς μπορεί να δοθεί ένα προστατευτικό καθεστώς σε ένα πρόσωπο που δεν γνωρίζουμε ποιο είναι, μη εντοπισμένο. Τώρα, σχετικά με τις ανώνυμες καταγγελίες, εγώ δεν λέω ότι δεν αντιμετωπίζονται, ίσα ίσα για τις επιχειρήσεις μπορεί να είναι ένα μέσο, θα έλεγα, που χρησιμοποιείται μη συμβατό με κάποιες βέβαια νομικές ρυθμίσεις. Σε πολλές περιπτώσεις ξεκινούν εσωτερικές διοικητικές έρευνες, αλλά στα πλαίσια του καθεστώτος δεν είναι κάτι που εντάσσεται στα πλαίσια του καθεστώτος προστασίας του καταγγέλλοντος. Σχετικά με το βάρος της απόδειξης, αυτή τη στιγμή κάνει ανάλυση μια, μια εταιρεία, μια ανάλυση της καταγγελίας, τότε χρησιμοποιεί συγκεκριμένες έννοιες και όρους έτσι ώστε να προχωρήσει στην καλύτερη δυνατή ανάλυση της καταγγελίας. Τώρα σε ένα θέμα στο οποίο δεν ήρθα, δεν μίλησα προηγουμένως και πρέπει να επανέλθω. Τώρα είχα πει ότι είμαστε υπέρ έτσι ώστε το πεδίο θα έλεγα των καταγγελιών να είναι κάτι που άπτεται των εθνικών και ευρωπαϊκών ρυθμίσεων. Τώρα, η προστασία του γενικού συμφέροντος ή η απειλή εις βάρος του γενικού συμφέροντος ε, για τις επιχειρήσεις. Τι γίνεται τώρα, όταν πάρει μια καταγγελία μια επιχείρηση, ξεκινά μια εσωτερική διαδικασία έρευνας, ίσως και με εξωτερική βοήθεια, και μετά αφού ολοκληρωθεί θα στραφεί στη δημόσια διοίκηση, στις δημόσιες αρχές και ίσως ε, να καταθέσει μηνύσεις κτλ. Το θέμα είναι πώς μπορεί να πάρει κάποια εσωτερικά μέτρα και να πάρει κάποιες κυρώσεις, να αποφασίσει κάποιες κυρώσεις μόνο με βάση μιας αρχής αρκετά θολής όπως αυτή του Γενικού Δημοσίου Συμφέροντος. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Λάγκεν τώρα και την Προεδρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, έπρεπε να πάω σε ψηφοφορία, αλλά δυστυχώς καθυστερήσαμε επειδή ο πρόεδρος είχε, ξεχάσει τα γυαλιά του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Τόμας Μαν έχει το λόγο. Όχι, α, Α, διαδικασία Catch Άννα Γκόμες. Και η, η κυρία Βέντερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πράγματι να επιβεβαιώσω ότι όσον αφορά τους καταγγέλλοντες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι σημαντικό να μπορεί κανείς να προσφύγει στον Όλαφ. Υπάρχει μία υπόθεση μιας ε, κυρίας που έχει αποκαλύψει κάποια συστήματα εκβιασμού των ε, κρατών μελών που σε αυτή την περίπτωση έχει οδηγήσει σε άλλη αντίδραση την Ευρωπαϊκή, από τον εργοδότη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην αρχή θεωρήθηκε ε, ενώ τώρα φαίνεται να είναι θέμα εκβιασμού. Ε, για να πληρώσει τις μέρες ε, που, ε, που δεν εργάστηκε. Θα ήταν ενδιαφέρον να οργανώσουμε σχετική ακρόαση. Η ερώτησή μου είναι, δεν θα έπρεπε να θεωρήσουμε ότι θα πρέπει να είναι αιτία παροχής ασύλου η καταγγελία παρατυπιών σε τρίτες χώρες. Δηλαδή κάποιος που καταγγέλει παρατυπίες ε, συχνά ε, βλέπει να παραβιάζονται τα ανθρώπινα του δικαιώματα. Μήπως θα έπρεπε αυτό να είναι αιτία παροχής ασύλου. Σας ευχαριστώ. Ε, δύο ερωτήσεις θα ακούσουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να επανέλθω στο θέμα του ορισμού. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι η προστασία των καταγγελόντων θα πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία, την ποιότητα των πληροφοριών. Ε, νομίζω όμως ότι αυτό ακριβώς ε, εννοούσε η ένα, Ο καταγγέλων κάνει κάποιο λάθος, πιστεύοντας ότι οι πληροφορίες που καταγγέλει πληρούν τα αντικειμενικά κριτήρια, διαπιστωθεί όμως ότι δεν τα πληρούν. Ε, από τις απαντήσεις σας ε, κατάλαβα ότι η καλή πίστη δεν ε, αρκεί διότι έχει να κάνει με την πρόθεση ενώ εμείς θα πρέπει να μιλάμε για αντικειμενικά κριτήρια. Και δεύτερον, όσον αφορά τα αντικειμενικά κριτήρια και τον ορισμό τους. Ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουμε πάντα να προστατεύουμε κατακέλλοντες που αποκαλύπτουν πληροφορίες ε, νόμιμα. Ε, είχαμε την ίδια συζήτηση όσον αφορά το εμπορικό απόρριτο. Εξετάσαμε περιπτώσεις καταγγελιών. Για παράδειγμα, οι αποκαλύψεις του Edward Snowden σίγουρα ήταν κρίσιμες για την ε, βελτίωση του κανονισμού για την προστασία δεδομένων. Ε, μπορεί λοιπόν ε, να έχουμε αποκάλυψη νομίμων πρακτικών που να πρέπει όμως να οδηγήσουν σε τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε να καθιστούν παράνομες. Είδαμε λοιπόν αρκετή σύγχυση ιδιαίτερα όσον αφορά την μετάφραση του όρου wrongdoing, πόσο μάλλον που ο δικαστής στην περίπτωση LuxLeaks χρησιμοποιούσε διαφορετική γαλλική μετάφραση του όρου αυτού από ότι το κοινοβούλιο. Το θέμα του wrongdoing, λοιπόν, είναι, θεωρείται ε, ότι πρέπει να έχει γίνει κακή πρακτική, ε, καλύπτεται η καλύπτονται οι παράνομες ενέργειες, ε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη αυτή ή να επικεντρωθούμε αποκλειστικά στο δημόσιο συμφέρον ε, και έναν ενδεικτικό κατάλογο. Πώς ε, θα πρέπει να διατυπώσουμε τον κανόνα ώστε να φροντίσουμε να καλύπτονται οι καταγγέλλοντες παρατυπίες που πρέπει να καλύπτονται. Ευχαριστώ. Ε, ναι, πολύ ευχαριστώ θα απαντήσω σε αυτό. Νομίζω ότι ο ενδεικτικό κατάλογο ε, θα είναι η απάντηση. Διότι πάντα θα υπάρχουν γκρίζε ζώνε στο θέμα αυτό. Ε, το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, λέει ότι οποιοδήποτε κάνει, ε, διαπράττει κάποιο αδίκημα ε, θα πρέπει να τιμωρείται. Ε, η ε, ανεξιθρησκεία, για παράδειγμα, δεν ήταν νομική υποχρέωση Θεωρήθηκε όμως ότι η... μάλλον ε, ε, στο παρελθόν δεν ε, προστατευόταν απαραίτητα κάποιος κατά των διακρίσεων λόγω θρησκείας. Χρειαζόμαστε ενδεικτικό κατάλογο και νομίζω ότι ο σχετικός Ιρλανδικός νόμος είναι καλός που περιλαμβάνει αυτά που περιλαμβάνει και ο αντίστοιχος νόμος του Ηνωμένου Βασιλείου, περιλαμβάνει όμως και κατηγορίες ή παραδείγματα από το αμερικανικό δίκαιο, όπως είναι για παράδειγμα η κακή διαχείριση. Θα υπάρχουν λοιπόν πάντα γκρίζες ζώνες. Νομίζω όμως ότι πολλά από τα θέματα αυτά έχουν καλυφθεί στη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, και τις κατευθυντήρες γραμμές ε, που το συνόδευαν. Όσον αφορά την πώληση των πληροφοριών που νομίζω ότι κάποιος ανέφερε, στο δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου, εάν ωφελείται κανείς προσωπικά από την αποκάλυψη, όταν αποκαλύπτει κανείς κάτι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν προστατεύεται. Είναι λοιπόν πολύ πιο εύκολο να προστατεύεται κανείς εάν αποκαλύψει κάτι εσωτερικά. Ε, λίγο πιο πολύπλοκα είναι τα θέματα εάν ε, προσφύγει κανείς σε κάποια αρχή. Εάν όμως η αποκάλυψη είναι πιο ευρεία, ε, τότε εξετάζεται εάν εάν πουλήσει κανείς την ιστορία του, για παράδειγμα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι θεωρείται αυτό επαρκής αποζημίωση. Όταν λοιπόν έχουμε ευρεία αποκάλυψη είναι πολύ πιο δύσκολη η προστασία διότι ε, αντισταθμίζεται το δημόσιο συμφέρον. Θα πρέπει όμως ε, να υπάρχει η ευελιξία, να μπορεί κανείς να απευθυνθεί κανείς απευθείας στα μέσα ενημέρωσης, αν αυτό είναι απαραίτητο. Ε, θα πρέπει να έχει την επιλογή να μην αποκαλύψει κανείς κάτι εσωτερικά προτού προσφύγει σε άλλους ε, τομείς. Ευχαριστώ. Να πω στην κυρία Γκόμες, ευχαριστώ που επαναφέρατε την προσοχή μας στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εμείς ενημερώσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μιλήσαμε με τους αρμόδιους υπαλλήλους. Επανέρχομαι σε αυτά τα οποία υπόθηκαν σε μια πρώτη φάση θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι καταγγέλλοντες χαρακτηρίζονται από αυτό που ονομάζουμε δημόσιο συμφέρον. Το ότι η συγκεκριμένη καταγγελία και η δημοσιοποίηση κάποιων προσπαθειών διάκρισης ανάμεσα σε μια καταγγελία δημοσίου συμφέροντος από τη μία και σε μια διαρροή πληροφορίας από την άλλη, είναι κάτι το οποίο ε, θα έλεγα δεν έχει ιδιαίτερη βάση λόγω ακριβώς της ιδέας, της ιδέας του δημοσίου συμφέροντος που φύγεται από συμπεριφορές διοικητικές κτλ. Τώρα για τις πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις σε σχέση με τα λεγόμενα αντικειμενικά κριτήρια. Το θέμα της regulations and because of different legal systems, there are legal systems in member states that are much more open. For example, not, not even just that there is the, the, the act has already been. Το θέμα, εν πάση περιπτώσει, των ανάρμοστων, όπως λέει η συνάδελφος πράξεων, είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο να ορίσει κανείς και είναι δύσκολο να ληφθεί υπόψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο καταγγέλων δεν έχει σαν στόχο το να καταγγείλει άπαξ κάτι, αλλά ο εργαζόμενος το άτομο να μπορεί να καταγγείλει κάτι ακόταν και όταν υποπτεύεται ότι κάτι μπορεί να συμβεί. Και γι' αυτό εγώ συμμερίζομαι με την κατηγοριοποίηση αυτή εν μέρη μόνο, γιατί τελικά ακόμα και οι καλύτεροι νόμοι δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις περιπτώσεις που μπορεί να εμφανιστούν. Το να είναι κανείς λεπτομερής και επακριβής είναι κάτι το οποίο μπορεί θα έλεγα να είναι αντίθετο με την ιδέα ότι θα υπάρξει περισσότερη κατανόηση και ευκρίνεια. Γι' αυτό λοιπόν το λεγόμενο wrongdoing είναι κάτι το οποίο δίνει κάποιες δυνατότητες, αλλά δεν είναι θα έλεγα μία ξεκαθαρισμένη έννοια, απλά αφήνει κάποια δυνατότητα περιγραφής μιας κατάστασης και στο τέλος στην ουσία δίνει την δυνατότητα να φτάσει μια διαδικασία στα δικαστήρια. Οπότε εκεί θα αποφασίσει το δικαστήριο όταν έχουμε να κάνουμε με μια υπόθεση προστασίας δημοσίου συμφέροντος ή όχι. Ε, και υπάρχει μια κάποια, ένα κάποιο επίπεδο μη προβλεψιμότητας. Πάντως καλύτερα να ε, είναι ανοιχτό το πεδίο και να μην είναι κανείς απόλυτος αποκλείοντας κάποιες δράσεις που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν την δημόσια αποκάλυψη κάποιων γεγονότων. Θα συμφωνήσω με την παρακαθήμενη συνάδελφο για τον χρονισμό και τις προθεσμίες ε, είναι πολύ σημαντικό πράγμα και όπως είπε και η συνάδελφος πολλές φορές δεν είναι τμήμα των κριτηρίων τα οποία καθορίζονται. Ποιος είναι ο βασικός στόχος, εν πάση περιπτώσει, είναι η διαδικασία για τον καταγγέλλοντα να παίρνει κάποιες πληροφορίες και να χρησιμοποιεί μια διαδικασία η οποία να επιτρέπει την αξιολόγηση της καταγγελίας και όχι μόνο απλά να γίνεται η καταγγελία, να ασχολούμεθα με τον καταγγέλλοντα και να ξεχνάμε το περιεχόμενο της καταγγελίας. Πρέπει να είμαστε πιο σαφείς εδώ λέγοντας ότι αν εμένουμε κυρίως στην καλή πίστη και στα προσωπικά στοιχεία και χαρακτηριστικά τότε η διαδικασία θα έλεγα κολλάει στην αρχική φάση και δεν επιτρέπει μια εξελεκτική διαδικασία η οποία να επιτρέπει την πραγματική αξιολόγηση της κατάστασης. Μια τελευταία σύντομη ερώτηση. Ένα λεπτό παρακαλώ. Κρέσπο. Σύντομα. Δεν μου δώσατε απάντηση για το πώς μπορεί η οδηγία για το εμπορικό απόρριτο, την οποία ενέκρινε το Κοινοβούλιο μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πώς θα μπορούσε να παρεμποδίσει την προστασία των καταγγελόντων στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα. Και μια δεύτερη ερώτηση. Στην Επιτροπή ΕΚΟΝΤ νομίζω έχουν ε, γίνει κάποιες προτάσεις και μέτρα ε, για το ανεξάρτητο σώμα συλλογή των πληροφοριών, μια ε, οντότητα, μια υπηρεσία ειδική στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου για να συλλέγει τις πληροφορίες των καταγγελόντων και πώς μπορούν να καθοριστούν στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποια δίκτυα επικοινωνίας, κάποιοι δίευλοι επικοινωνίας, δημιουργώντας ένα πρωτόκολλο έτσι για την λειτουργία των διαδικασιών καταγγελίας. σχετικά με το εμπορικό απόρριτο, επιχειρηματικό απόρριτο. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι το οποίο απαγορεύει την προστασία των καταγγελόντων για δημόσιους λόγους, για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Στην οδηγία αυτή πράγματι, αν θέλετε, η βασική αντίληψη είναι η προστασία ε, του απόρριτου ακόμα και των καταγγελόντων δεν παρεμποδίζει λοιπόν την προστασία τους. Αυτό το οποίο έχει σημασία και έρχομαι εδώ στις ερωτήσεις οι οποίες τέθηκαν για τα λεγόμενα αντικειμενικά στοιχεία της καταγγελίας, νομίζω ότι ε, πρέπει να περάσουμε στην ευρύτερη δυνατή προσπάθεια ορισμού της καταγγελίας για λόγους δημοσίου συμφέροντος, κάτι το οποίο θα επιτρέψει να αποφύγουμε στο να μείνουμε σε ένα σαφές επίπεδο αποκλειστικά καταγγελτικό. Και ο ορισμός αυτός θα πρέπει να συνοδεύεται με αυτήν την βαθμιαία προστασία, με αυτούς τους διάβλους ε, ε, καταγγελίας, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη τα συμφέροντα της επιχείρησης και τα συμφέροντα της κοινωνίας, η οποία θα πρέπει ακριβώς να μπορεί να αντιδρά και αυτή η προσπάθεια εξισορρόπησης των συμφερόντων είναι κάτι το οποίο ξεπερνά την συγκεκριμένη οδηγία. Ευχαριστώ. Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι? 30 δευτερόλεπτα. Να πω απλώς ότι η οδηγία αυτή όντως ήταν ενισχυτική και σε ό,τι αφορά τις διαρροές των ε, ε, πληροφοριών είναι το, ε, όταν γίνονται διαβρώσεις πληροφοριών είναι τότε που αρχίζουν να καταπατώνται τα στοιχεία της ε, εμπιστευτικότητας Δεν μπορεί να κρύψει κανείς την κακοδιαχείριση επειδή υπάρχει εμπιστευτικότητα. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται αυτό για να κρυφτεί μια κακοδιαχείριση. Και αυτό πρέπει να τονίσουμε εδώ. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και τις πέντε εμπειρογνώμονες. Πολύ ενημερωτικά αυτά που μας είπατε. Μόνο γυναίκες είχαμε σήμερα στην ε, Επιτροπή μας. Πολύ ε, ενθαρρυντικό. Έχουμε την, ε, τον κύριο Γέτσεκ, την κυρία Γκροσιά και τον τρίτο συνεισηγητή για την σχετική έκθεση. Ευχαριστώ τον συμπρόεδρο, τον κύριο Σβόποντα. Συζητήσαμε δύο ώρες και δύο λεπτά. Ε, και νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε τώρα τη συνεδρίαση. Okay.